le train de Paris était à l'heure. Guten Morgen, guten Morgen, morning. Πολύ καλημέρα σας, καλημέρα σε διάφορες γλώσσες, καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα έχουμε μια πρωία με πολλές ψηφοφορίες και σημαντικά θέματα φυσικά στην ημερήσια διάταξη. Καλωσορίζω λοιπόν όλους θερμά στη συνεδρίασή μας και έχουμε και όσο δεν είμαστε όσοι και χθε, αλλά παρόλα αυτά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και μια πρόταση τώρα για την τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης που έχει υποβληθεί. Η κυρία Ροβάνα έχει ζητήσει την δική της τροπολογία να την ψηφίσουμε μετά την πρώτη, μετά την 112, το σημείο 13 της ημερησίας διάταξης διότι πρέπει να πάει να παρουσιάσει μια άλλη εισήγηση. Αν δεν υπάρχει ένσταση, ξεκινάμε με το σημείο 7 στην ημερήσια διάταξη. Μετά 13 και μετά θα συνεχίσουμε με το 8, 9, 10 και τα λοιπά. Συμφωνείτε, δεν υπάρχει κάποια ένσταση, βλέπω. Και θα βοηθήσουμε να εργαστεί και στην άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή συνάδελφο. Αυτό είναι καλό. Όλοι έχετε τι κάρτε για την ψηφοφορία σήμερα. Θα υπάρξουν και με ονομαστική κλίση ψηφοφορίε. Αν δεν τις έχετε να πάτε να τις φέρετε γρήγορα γιατί θα χρειαστείτε τις κάρτες σας. Ένα μικρό λεπτό δώστε μου. Λοιπόν, 7 καθολικές υπηρεσίες εισηγητής είναι ο Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες. Περνάμε αμέσως στην ψήφιση. Τροπολογία 1, τάκουλα, υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 3, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 4, υπέρ. Κατά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 κατά αποχές εγκρίθηκε 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 21 υπέρ κατά αποχές και αυτή εγκρίθηκε 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 26 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 56 υπέρ. ένα εναντίον, καμία αποχή. Θερμά συγχαρητήρια στον εισηγητή Φερνάντες. Συγχαρητήρια για την 112 για τις υπηρεσίες που θα βοηθήσει πολλούς στην Ευρώπη να έχουμε το 112 που μπορούμε να καλέσουμε σε περίπτωση ανάγκης. Και όπως είπαμε, Περνάμε αμέσως στο σημείο 13 της ημερησίας διάταξης. Προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδομή για το, μέχρι το 2020 και μετέπειτα. Συντάκτρια της γνωμοδότησης η κυρία Ροβάνα Λαμ. Περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. <clears throat> Γεμπράντι. Όχι, όχι ακόμη. Τι συμβαίνει, παρακαλώ. το ΕΛΚ θα διανύμει τον πίνακα ψηφοφορίας. Να περιμένουμε λοιπόν πρώτα να γίνει και αυτό. Πολύ καλά. Λοιπόν, ανταλλαγή των πινάκων ψηφοφορία μεταξύ κοινοβουλευτικών ομάδων που πρέπει να γίνει. Εν τω μεταξύ και ο συνάδελφος Σνέρχαρτ πήρε και τον πίνακα ψηφοφορία. Πολύ καλά. Σνέρχαρτ. Βρίσκεται εδώ, όχι. Ακόμα όχι. Έστω. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται έχουν όλοι πάρει τους πίνακες για την ψηφοφορία, τους κατάλογους και μπορούμε έτσι φυσικά να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ξαναξεκινάμε, τροπολογία 1, <clears throat> Γεμπράντι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε, 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε ή 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 6 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 9 8 να ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία 8 από το ΕΛΚΑ ένας παραπάνω που συμμετείχε στην ψηφοφορία όλα εντάξει πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε η 8 απορρίφθηκε η εννέα τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Η δέκα, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. δέκα. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 22 υπέρ κατά α, αποχές απορρίφθηκε ναι έλεγχος εντάξει ψηφίζουμε την 22 άρχεται η ψηφοφορία Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Απορρίφθηκε μάλιστα. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 27 αλφα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 29 υπέρ κατά αποχές και αυτή εγκρίθηκε 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και τώρα φτάσαμε ήδη στην τελική ψηφοφορία πια για αυτή την έκθεση άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά Τέλος ψηφοφορίας. 56 υπέρ. 3 εναντίον, μία αποχή. Θερμά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια Ροβάνα Πλάμπ. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ε, ψήφιση προς έγκριση για και ευχαριστούμε και τη Γραμματεία για αυτό, την, την προετοιμασία των πινάκων ψηφοφορίας και που έκανε πολύ καλή δουλειά από τη Γραμματεία πριν από την ψηφοφορία. Συνεχίζουμε λοιπόν με το σημείο 8 στη συνέχεια. Και ε, την ψήφιση για την δική μας έκθεση εκπομπή ρήπων πέραν των 20% και τον εκτίμηση κινδύνου διαρροής άνθρακα. Η συγητής ε, Has äh, Μάλιστα. Έχουμε τροπολογία για ονομαστική κλίση ψηφοφορίες με ονομαστική κλίση. Γίνεται αυτό με βάση τον κανονισμό στην δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπή σε σχέση με τις τροπολογίες 2 και 2α λοιπόν. Και πρέπει να ρωτήσω αν κάποιος έχει ένσταση να κάνουμε ονομαστικές ψηφοφορίες. Πρέπει το αντίστροφο τώρα να γίνει. Ένα τέταρτο των μελών, 16 μέλη πρέπει να καταμετρηθούν που θέλουν την ονομαστική ψηφοφορία. Λοιπόν, όσοι την επιθυμούν να ηγερθούν. Φαίνεται ότι είναι πάνω από 16, είναι σαφές, γίνεται δεκτή ονομαστική ψηφοφορία. Πολύ καλά. Και θα γίνει η ονομαστική ψηφοφορία. Και ξεκινάμε με τον συμβιβασμό 1. Ποιοι είναι υπέρ του συμβιβασμού 1. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός υπαριθμών 2. Είναι η ονομαστική ψηφοφορία τώρα αυτή. Ονομαστική, με ονομαστική κλίση ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. 53 υπέρ 7 εναντίον. Μία αποχή. Έγινε δεκτή αυτή η τροπολογία. Και περνάμε στην ολοκληρωμένη τροπολογία 1. Πάγια τροπολογία 1. Αυτόν τι είναι τώρα το 2α, αυτή είναι η 2α. Πάλι με ονομαστική κλίση λοιπόν ψηφοφορία και για αυτή την ολοκληρωμένη ψηφο, ε, τροπολογία άρχεται η ψηφοφορία μας ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 36 υπέρ 27 εναντίον. Καμία αποχή εγκρίθηκε. Περνάμε στον συμβιβασμό 3 τώρα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Συμβασμό 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμό 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμό 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμό 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 14 υπέρ παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 15 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε. 16 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε. 17 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε. 18 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε. 19 υπέρ κατά αποχές και αυτή εγκρίθηκε. Τώρα αυτό διευκολύνει φυσικά το έργο και πολύ μάλιστα. Πάμε πίσω πολλές σελίδες τώρα διότι δόξα τω Θεώ είχαμε τόσες πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες. Σε μένα είναι τώρα η σελίδα 11 εκεί που συνεχίζουμε. Σωστό. Εν πάση περιπτώσει. Παράγραφος 2α νέα. Τροπολογία 98 λοιπόν. Σαμπίνε Βίλς η συντάκτρια. Και έχουμε σε τμήματα ψήφιση. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Α, καταπίπτει. Μάλιστα, το δεύτερο καταπίπτει. Συνεχίζουμε με την τροπολογία 101. Ορέστε Ρώση υπέρ. Κατά απόχες απορρίφθηκε 102 υπέρ κατά απόχες απορρίφθηκε 103 υπέρ κατά απόχες απορρίφθηκε 104 υπέρ κατά απόχες έλεγχος ψηφίζουμε την 104 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά Ένας από το ΕΛΚ που ψηφίζει και είναι παραπάνω. Εντάξει, πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα, απορρίφθηκε. 27 υπέρ 34 εναντίον απορρίφθηκε. 105 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Η 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η 108 σε αρκετά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και τώρα τι κάνουμε τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές και αυτό εγκρίθηκε 109 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε επόμενη σελίδα τώρα παράγραφος 5α 118 τροπολογία σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές και αυτό απορρίφθηκε. Συνεχίζουμε. Παράγραφος 5α νέα, 121 τροπολογία, Westland. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Ταυτόσημη 122 και 123 υπέρ αυτών. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκαν. Περνάμε στην 126 υπέρ κατά αποχές. Θα, θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν αυτή την τροπολογία. Πέρας ψηφοφορίας. Λοιπόν, με πολύ μικρή διαφορά απορρίφθηκε. 124 υπέρ. Κατά. Και εδώ πρέπει να ελέγξουμε την 124. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα Τώρα είναι αντίστροφο το αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε με μικρή διαφορά. Εγκρίθηκε. Δύο συνάδελφοι όμω δεν έχουν κάρτα ψηφοφορία. Και γι' αυτό δεν ξέρουμε την ακρίβεια του αποτέλεσμα. Σε πάση περιπτώσει, 125 καταπίπτει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 131 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 136 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 136 άρχεται η ψηφοφορία ένας από το ΕΛΚ παραπάνω εξακολουθεί ένας παραπάνω από το ΕΛΚ ναι εντάξει πέρας ψηφοφορίας τώρα λοιπόν απορρίφθηκε το αποτέλεσμα 135 σε διάφορα τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά έλεγχος. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της 135 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ. Καταπίπτει λέτε, ναι. Μάλιστα. Αν δεν εγκριθεί, λέει, καταπίπτει το δεύτερο τμήμα, πάει αυτό. Και μετά η 134 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Η 132 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Μετά το δεύτερο τμήμα της 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε αυτό. Μετά 137 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 138 να το ελέγξει ο, ο 137 άρχεται η ψηφοφορία τώρα πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε μετά έχουμε την 138 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 140 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 142 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 143 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 143 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα Πρέπει να επαναλάβουμε δυστυχώς, διότι το τελευταίο δευτερόλεπτο είχαμε ένα από το ΕΛΚ παραπάνω που συμμετείχε. Λοιπόν, άρχεται και πάλι η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Είσαστε άτυχοι, ωραίο θα ήταν. Και πάλι ένας από το ΕΛΚ παραπάνω. Τώρα είναι τα πράγματα εντάξει, αλλά παραμένει σε ισοψηφία το αποτέλεσμα, δηλαδή απορρίφθηκε η τροπολογία. Εντάξει. Πάμε στην 144, Φρανσουάς Γκροστέτ, υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίθηκε, 145, υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίθηκε, 100... 46 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 149 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 148 σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε καταπίπτει το δεύτερο μια και απορρίφθηκε το πρώτο η 147 τώρα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίθηκε. Η 150 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίθηκε. 100. 52 καταπίπτει 151 πρώτο τμήμα κατά αποχές απορρίφθηκε. Μετά πάμε στην 153 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συνεχίζουμε με την παράγραφο 10α. Νέα 164 τροπολογία και 165 υπέρ αυτών των δύο. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. Έλεγχος. Εντάξει. Ψηφίζουμε την 164 και 165 ηλεκτρονικά. Έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκαν. Η 166 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Η 167 με προφορική τροποποίηση, υπέρ, κατά, αποχές, Δεν είναι σαφέ το αποτέλεσμα. Δεν είδα του φιλελεύθερου. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε αυτή την τροπολογία 167 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ένας από το ΕΛΤ παραπάνω που συμμετέχει. Τώρα τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 168 τώρα υπέρ Α, επειδή απορρίφθηκε λοιπόν, επανερχόμαστε στο αρχικό κείμενο της 167, αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τώρα, ναι, να ελέγξουμε λέτε, ηλεκτρονικά. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα, ναι, απορρίφθηκε λοιπόν. Πάει, εντάξει. Δεν βλέπουμε και όλοι με τέτοια σαφήνεια τα χέρια. Τέλος πάντων, 168 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Ήτρε 1 είναι υπέρ ήτρε 1. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Ήτρε 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Ήτρε 4. Ήτρε 3 διορθώνει ο πρόεδρος υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Ήτρε 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και τώρα ήτρε 6 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας Αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε. Τώρα συνεχίζουμε. Χαιρετίζω και την εισηγήτρια Ήτρε Ρωμάνα. Είσαστε εισηγήτρια, έτσι δεν είναι, για αυτή την έκθεση. Εντάξει, συνεχίζουμε με την τροπολογία 220 υπέρ. 220 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Στη συνέχεια 220 θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 220. Τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Τρεις που δεν συμμετέχουν. Και όταν γίνεται αυτό, είναι πολύ στενό το αποτέλεσμα, απορριφθείται 9, λοιπόν, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Είτε 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ήτρε 17 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 169 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 170 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 171 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Συνεχίζουμε με την τροπολογία 173 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 174 σε τρία τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε να ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε το δεύτερο της 174, άρχεται. Ένας από το ΕΚ παραπάνω στην ψηφοφορία, δύο παραπάνω τώρα. Τώρα εντάξει. Λοιπόν, τέλος ψηφοφορίας τώρα και ισοψηφία 31-31. Με μία αποχή. Απορρίφθηκε. Μάλιστα. Περνάμε στην 175 τώρα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε τρίτο τμήμα υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 177 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ ακαταπίπτει το δεύτερο τμήμα πολύ καλά και το τρίτο πάει και αυτό 178 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 179 υπέρ κατά αποχές και αυτό εγκρίθηκε 180 δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία ένας από το εκ παραπάνω. Είσαστε πάρα πολύ, θα έλεγα, επιμελή σήμερα το πρωί, με ιδιαίτερο ζήλο. Απορρίφθηκε το αποτέλεσμα. 181 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 183 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Και τώρα 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 185 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 186-187 ταυτόσημες υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν 188 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ α καταπίπτει αυτό πολύ καλά καταπίπτει Εκατόν υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Ήτρε 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ήτρε 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 197 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε ήτρε 36 έλεγχος λέτε εντάξει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 197 άρχεται η ψηφοφορία μας ένας από το εκ παραπάνω και πρέπει να αποσαφινιστεί τώρα αυτό απορρίφθηκε 197. Η Φρανσουάς Γκροστέτ είχε καλό μάτι σήμερα ελέγχοντας τα πράγματα. Και έτσι πάνε καλά τα πράγματα. Εντάξει, λοιπόν, ήτρε 36. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 198 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 199 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 202 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 206 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 207 ε, υπέρ κατά αποχές, έλεγχος, ψηφίζουμε την 207 ηλεκτρονικά, άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Ist Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Geht es mit Συνεχίζουμε με την παράγραφο 16α νέα τροπολογία 217 ή τι λέτε Παράγραφος 17α, 229, υπέρ της 229. Κατά αποχές εγκρίθηκε. ήτε 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 230 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές και αυτό εγκρίθηκε 231 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 232 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 233 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 200 34 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές και αυτό εγκρίθηκε Δεύτερο τμήμα. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, έρχεται η ψηφοφορία. Από το ΕΛΚ και πάλι παραπάνω, εντάξει, τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα αυτή τη φορά ήταν σωστό. Εγκρίθηκε. 235 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 237 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 203-204 ταυτόσιμες υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 228 328 διορθώνει ο πρόεδρος υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 238 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 239 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 241 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 243 υπέρ 242 διορθώνε πρόεδρος υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 200 Έλεγχος ζητείτε. Λοιπόν, να ελέγξουμε, έστω. Ψηφίζουμε την 242 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Θα λέγα εγκρίθηκε. Λοιπόν, αφού είναι σαφές πλέον, μπορούμε να πούμε πέρας ψηφοφορίας είτε με το πράσινο είτε το κόκκινο εγκρίθηκε τέλος πάντων μάλιστα που είχαμε σταματήσει 40. Τώρα έχουμε τη ΣΥΤΡΕ την 30 και την 243 υπέρ. Α, είμαστε 242, 243 τώρα. Holger Kramer υπέρ. κατά έλεγχος ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 243. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Και τώρα αυτή εγκρίθηκε μάλιστα. 244 και ήτρε 30 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκαν. 245 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 246 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 247 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 248 καταπίπτει αυτή 249 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Να ελέγξουμε, θέλετε. Να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 249 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορία και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 251 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 252 και 253 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 21 υπέρ Ήτρε 19 διορθώνει ο πρόεδρος Ήτρε 19 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 21 υπέρ κατά άποχες και αυτή εγκρίθηκε Ήτρα 28 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε Ήτρα 29 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε. Ήτρε 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Ήτρε 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Ήτρε 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Είτε 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η τροπολογία 117. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Μάλιστα, έχουμε την Ήτρε 38, πρώτο τμήμα, να ψηφίσουμε υπέρ. 38, πρώτο, 138 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, Δεν είναι πλέον σαφές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ή 38. Από το ΕΛΚ ένας παραπάνω στην ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν. Είναι σαφέστατο το αποτέλεσμα. Απόλυτα σαφές. Αλλά δεν σηκώνονται τα χέρια. Τέλος πάντων, η 117, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Μετά 254 Να ελέγξουμε λέτε λοιπόν, ωραία, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 117 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πρώτο τμήμα, άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε με το δεύτερο τμήμα φυσικά. Ποιοι είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος κατά αποχές και αυτό εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 254 υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε 255 υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε 257 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε ήτρε Y342. υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε ήτρε Y344. υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 259 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 260 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το πρώτο τμήμα της 260 τέλος ψηφοφορίας αποτέλεσμα απορρίφθηκε 261 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τι λέτε έλεγχος να ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν τέλος ψηφοφορίας εγκρίθηκε μια σειρά συναδέφων όμως δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Λοιπόν, εγκρίθηκε έστω. 262 τώρα, υπέρ. Κατά. Απόχες. Και εδώ θα πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία πάλι. Από το ΕΛΚ ένας παραπάνω. Τώρα εντάξει και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 263 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Ήτρε 41 υπέρ. Κατά δεν μπορώ να αναγνωρίσω ποιο είναι το αποτέλεσμα με τα χέρια σας και πάλι 41 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε 273 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε παράγραφος 21α νέα 284 τροπολογία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε θα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα άρχεται Τέλος, εγκρίθηκε. Κύριοι, πρέπει να σηκώνετε τα χέρια σας, να βλέπουμε τι γίνεται. Κανένας δεν σηκώνει τα χέρια και πρέπει να μπορώ να βλέπω ως πρόεδρος πώς ψηφίστε. Δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ του δευτέρου τμήματος. Κατά άποχες εγκρίθηκε. 285 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 286 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε να ελέγξουμε εντάξει 286 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται πέρας εγκρίθηκε 293 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 294 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 295 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 296-297 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν ψηφίζουμε επ' αυτών άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά τέλος ψηφοφορίας απορρίφθηκαν. 298 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Ήτρε 40 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην παράγραφο 26α νέα, τροπολογία 318, αϊκότ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Περνάμε στην 320, υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 321 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 323 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 323 Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 322 τώρα, υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 322. Άρχεται ist angenommen. Εγκρίθηκε. Φτάνουμε τώρα στην 326. Holger Kramer, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 326. Άρχεται. Τέλο Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε. 327 υπέρ. Κατά. Περίπου τα ίδια, αλλά πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Απορρίφθηκε. 329 τώρα υπέρ. 329 τροπολογία. Κανείς υπέρ. Υπέρ είπαμε. Λοιπόν, κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 320 υπέρ. 330 διορθώνει ο πρόεδρος. Μάλιστα. Υπέρ. Σωστό. 330 κατά άποχες εγκρίθηκε. 331 τώρα. Θα ελέγξουμε την 330. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά και άρχεται επί της 330. Τέλος ψηφοφορίας. Μάλιστα. Αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε. Έτσι. Πολύ καλά. 331 τώρα. Υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε Ήτρε 47 πρώτο τμήμα υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε Ήτρε 48 υπέρ κατά και πάλι επαναλαμβάνουμε ήτρε 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε επιτέλους ήτρε 49 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 300 και πάλι να ελέγξουμε εντάξει Φρανσουάζ έστω να ελέγξουμε τόσες πολλές φορές 339 τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αυτή τη φορά εγκρίθηκε αυτή. Τι να κάνουμε, εντάξει. Καταπίπτει επόμενη. 339-340 υπέρ αυτών. κατά αποχές απορρίφθηκαν. Το ξέρανε. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία έλεγχος επ' αυτών. 339-340. Τέλος ψηφοφορίας. Βλέπεις, να, αυτά συμβαίνουν καταψηφίστηκαν. Δεν έχουν όμως όλοι τις κάρτες, γιατί διαφορετικό αποτέλεσμα από τα χέρια που σηκώθηκαν πριν. Ψηφίζουμε την 341 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε, μάλιστα. 443 υπέρ. 343 διορθώνει ο πρόεδρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 344 υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Μάλιστα. Απορρίφθηκε. 345 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 346 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίζουμε την 346 άρχεται Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 347 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 51 ήτρε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 348 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 348. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Απορρίφθηκε. 349 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εδώ θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. «352 Γκαντίνι Μπερλάτο» με αρκετά σε τμήματα ψηφοφορίες. Πρώτο τμήμα υπέρ. Και αυτό καταπίπτει τι. Όλα. Μάλιστα. Πολύ καλά. 353 καταπίπτει και αυτή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 355 τροπολογία. Ρίτα κόρλα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 356 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 357 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές έλεγχος ωραία άρχεται ψηφίσατε όλοι Τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Μάλιστα. Αρχικό κείμενο. Ψηφίζουμε το αρχικό. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε το αρχικό κείμενο. Ήτρε 50. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την Ήτρε 50. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Τροπολογία 360 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 358 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε είπαμε. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, έλεγχος. Τι να κάνουμε. Άρχεται. Elle Ψηφίσατε όλοι, κάποιοι λείπουν ακόμα. Μάλιστα, τώρα εντάξει. Τέλος ψηφοφορές. εγκρίθηκε, συγχαρητήρια. Κέρσιο πριν. τι έκπληξη είναι αυτή. Ήτρε 52. τώρα ή τι λέτε. Καταπίπτει, ε. Μάλιστα. Πάει. Also, Amendment 359. 359 τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ της 359 παρακαλώ. Κατά άποχες. Εγκρίθηκε. Ήτρε 52 τώρα. Υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός έλεγχος ήτρε 52 άρχεται Υφίσατε <laughs> όλοι. Ναι, κάποιος άλλος. Εντάξει, τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα, απορρίφθηκε. Μάλιστα. 361 τροπολογία υπέρ. κατά, άποχες, έλεγχος και πάλι, άρχεται. Αιώνια θα διαρκέσει αυτό επιτέλους. Τι γίνεται. Τέλος ψηφοφορίας λοιπόν τώρα. Απορρίφθηκε. Ήτρε 53 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Ήτρε 54 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ήτρε 55 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ήτρε 56 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος, άρχεται. Τέλος πληροφορία, απορρίφθηκε. Ήτρε 57. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. Ήτρε 58. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. Ήτρε 59. Υπέρ. Κατά άποχες, απορρίφθηκε. Ήτρε 60, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίθηκε. Τροπολογία 362, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Πρώτο, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1 και 2 και 3 και 4. Ταυτόσημες υπέρ αυτών. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκαν. 5. Μόνο το δεύτερο τμήμα. Μόνο το δεύτερο τμήμα. Υπέρ του δεύτερου τμήματος. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Στι αιτιολογικέ σκέψει η τροπολογία 6. Έλεγχος, το δεύτερο τμήμα της 5. Πολύ καλά, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε μάλιστα. Λοιπόν, την επόμενη φορά να το σκέφτεστε πιο νωρί. Τι να κάνουμε. Τροπολογία 5 λέει ο πρόεδρο. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Διορθώνεται ο πρόεδρο. Α, όχι. Πάμε στην 6. Εκεί ψηφίζουμε. 6 και 7 ταυτόσιμε. Ψηφίζουμε αυτέ. Υπέρ αυτών. Κατά. Αποχέ. Εγκρίθηκαν. 8 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίθηκε. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 11 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 13 υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε 14 πρώτο τμήμα υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε 15 υπέρ κατά άποχες έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 16. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 18 Έλεγχος στην 17. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 19 υπέρ. κατά αποχές έλεγχος ψηφίζουμε την 19 άρχεται από το έλκενας παραπάνω τέλος ψηφοφορίας τώρα αποτέλεσμα απορρίφθηκε 20 υπέρ κατά Αποχές εγκρίθηκε. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Ήτρε αιτιολογική σκέψη Β υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 28 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. τοπολογία 29 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 30 η πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. 30 πρώτο τμήμα. Από τους Σοσιαλιστές και δημοκράτες ένας παραπάνω. Εντάξει τώρα. Τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Δεύτερο τμήμα της 30. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίζουμε το τρίτο τμήμα της 30. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Η ισοψηφία απορρίφθηκε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τροπολογία 39 και 40 σε αυτές τις δύο, υπέρ αυτών. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. Η επόμενη καταπίπτουν, οι επόμενες καταπίπτουν 42 λοιπόν τώρα. Εντάξει, 42 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Ψηφίζουμε την 42, άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Και απορρίφθηκε. 41 τώρα, υπέρ. Κατά, αποχές, έλεγχος. Ψηφίζουμε τη 41, άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα απορρίφθηκε και αυτή. Πάμε τώρα στην τροπολογία 51. Υπέρ. Υπέρ της 51. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 51 και άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας ε, για αυτή. Μάλιστα εγκρίθηκε το αποτέλεσμα. 52 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος και επ' αυτού. Πρώτο τμήμα της 52. Άρχεται. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Ε, τότε τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε λοιπόν. Η ισοψηφία απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα. Ναι. Δεν έχει νόημα. Καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. Πάμε στην Ήτρε. Στο recital A. Πρώτη αιτιολογική σκέψη. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε μετά στην τροπολογία 58. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 59 τώρα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 62 τροπολογία πρώτο τμήμα. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 65 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 66 υπέρ. 65 έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 65 λοιπόν. Τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε μάλιστα. Τροπολογία 66 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε 67 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικά ψηφίζουμε άρχεται 67 πρώτο τμήμα τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκε Και τώρα που πάμε. Τώρα πάμε στην τροπολογία 68. 68 λοιπόν. 68 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές και αυτό εγκρίθηκε μάλιστα καταπληκτικά και τώρα η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά από το ΕΛΚ ένας παραπάνω πάλι ψηφίσατε όλες και όλοι Τελ... Ψηφίσατε όλες και όλοι. Εντάξει, τέλος ψηφοφορίας τώρα. Αποτέλεσμα 44 υπέρ, 14 εναντίον, μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή Μπασάικοτ. Θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνατε και αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ όλους τις γραμματείας και όλους οι εισηγητές επίσης και συναδέλφους από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ήτρε για τη συνεργασία τους για το αποτέλεσμα αυτό στην έκθεση αυτή που θα υποβληθεί στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστούμε όλους και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε <clears throat> με τους ε, φρουτοχυμούς. Είναι το σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη αυτό. Λοιπόν. Σλούτερ, διαδικαστικό, παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω την, την νομική υπηρεσία της Επιτροπής να μας πούν τη γνώμη τους για τις συμβιβαστικές τροπολογίες 1 και 2. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλεγε ότι αν προσθέσει κανείς ζάχαρη σε ένα νέκταρ θα πρέπει αυτό να συμπληρωθεί δίπλα από το όνομα του προϊόντος. Αλλά το Κοινοβούλιο με αυτές τις κοινέ τροπολογίες αντιστρέφει αυτή τη λογική και λέει ότι δεν ε, αναφέρει την ζάχαρη όταν τη βάζεις παρά μόνο στα, στα, ε, στα στοιχεία τα οποία περιέχει το προϊόν. Αν ένας ε, χυμός φρούτου απαγορεύεται να έχει ζάχαρη Αναρωτιέμαι σε αυτή την περίπτωση αν έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις οδηγίες. Λοιπόν, ο εισηγητής έχει μια άποψη γι' αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η διάταξη αυτή συνεχίζει να υφίσταται για τους χυμούς που αποκαλούνται φυσικοί και για τους συμπυκνωμένους. Τα νέκτα εξορισμού δεν πρέπει να έχουν γλυκαντικέ ουσίε ή ζάχαρη. Δεν προσθέτουμε λοιπόν αυτή τη ζάχαρη είτε στου συμπυκνωμένους είτε στου αποκαλούμενου φυσικού χυμού. Επιτρέπουμε την προσθήκη ε, ζάχαρη ή γλυκαντικέ ε, ουσίε ή μόνο μέλι αποκλειστικά στα νέκταρ που εξ ορισμού πρέπει να έχουν αυτέ τι ουσίε. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό το οποίο αναφέρθηκε. Αυτή τη στιγμή ακόμα και χωρίς την, πρόσθετη, ε, την προσθήκη ζάχαρης μπορούν να έχουν 15 γραμμάρια για την οξύτητα καταπολέμηση αυτής. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος συμφωνεί με την άποψη του εισήγητη. Οι ομάδες ήταν όλες υπέρ, εκτός των πρασίνων. Γι' αυτό πρέπει να ψηφίσουμε. Λοιπόν, τροπολογία 21 τώρα. ρώτησα την Επιτροπή, όχι τον εισηγητή τι γίνεται. Βρισκόμαστε στη μέση ψηφοφορίας και ο πρόεδρος είναι υπέρ της άποψης ε, που παρουσιάστηκε και έτσι θα ψηφίσουμε σχετικά. Ακούσαμε τον εισηγητή τι είπε. Αυτό θα γίνει λοιπόν. Εν μέση ψηφοφορία δεν μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε συζητήσεις εκ νέου. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει εκ των προτέρων. Σνέρχατ που ζήτησε τον λόγο πιο πριν. Σύντομα, έχει δίκιο ο πρόεδρος. Πριν από την ψηφοφορία δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να αρχίσουμε με επιχειρήματα για αυτά. Όμως η ένσταση είναι νόμιμη, είναι θεμητή. Θα πρότεινα σε σχέση με την ψηφοφορία πριν την εξέταση στην Ολομέλεια αυτό το θέμα να το ξαναδούμε και πάλι, να το ξανασυζητήσουμε. Είναι εναντίον, θα ψηφίσουν εναντίον οι εναντίον. Είναι απλό. Δεν μπορούμε να ξαναρχίσουμε εδώ να συζητάμε τώρα εις το διηνεκές αν επιτρέπεται τέτοια προσθήκη ή όχι. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε. Όσοι είναι εναντίον μπορούν να καταψηφίσουν. Είναι απλό. Ορέστε Ρώση, τροπολογία 21, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 23, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Άγκρι, τι έχουμε, άγκρι 4, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία 24, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 25, υπέρ, κατά, αποχές, Έλεγχος. Ψηφίζουμε την τροπολογία αυτή είναι 25. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Λοιπόν, και περνάμε τώρα στις ολοκληρωμένες τροπολογίες. Στην περιβόητη 1 ολοκληρωμένη τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της Consolidated 1. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε στις Consolidated 2. Ποιοι είναι υπέρ της ολοκληρωμένης 2. Κατά άποχες εγκρίθηκε αυτή. Μετά πάμε στην Άγκρη 17 υπέρ. Άκρη, Άγκρη 7 διορθώνει ο πρόεδρος υπέρ. Κατά άποχες εγκρίθηκε. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 40 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε μετά δεύτερο τμήμα τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 41 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε άγριο 8 Άγριο 8 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Άγριο 9, υπέρ, τα αποχές εγκρίθηκε. Η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Άγκρη Γεωργίας 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Μετά πάμε στην τροπολογία 8. Τροπολογία 8 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε. 43 τροπολογία υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε. Άγκρι 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 46 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Πάμε στις 45 τώρα. Υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Άγκρι 13 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Άγκρι 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 10. Τοπολογία 10. Άγκρι 14. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Άγκρι 14. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Τροπολογία 10 και οι 44 ταυτόσιμες υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. Η 47 τροπολογία με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Άγκρι 16 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίθηκε. 50 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίφθηκε. 51 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Άγκρι 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 54 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίζουμε την 54. Άρχεται. Ένας από τους σοσιαλιστές παραπάνω. Τώρα εντάξει, τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Το αρχικό κείμενο αυτής της τροπολογίας 54. Ποιοι είναι υπέρ του αρχικού κειμένου της 54. 54 έτσι, αρχικό κείμενο υπέρ, χωρίς προφορική τροποποίηση. Ποιοι είναι υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε και στη συνέχεια τροπολογία 55 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε 56, 57, 58, 59 άγκρι 18 όλες ταυτόσιμες υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 60. Η 60 λοιπόν υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε. 61. Καταπίπτει, τι λέτε. Εξήντα υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε 62 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε άγκρι 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 63 υπέρ κατά άποχες. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την τροπολογία αυτή. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Άγκρι 20 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Άγκρι 21 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 64 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 13 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Άγκρι 22 υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε. Άγκρι 23 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Άγρι 24 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίθηκε. Άγρι 25 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίθηκε. Άγρι 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Η τροπολογία 16 με προφορική τροποποίηση. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Πάμε στην αρχική, στο αρχικό κείμενο της 16 υπέρ αυτού. Κατά αποχές και αυτό απορρίφθηκε. Και τώρα πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1 πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Η 17 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Άγρι 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Ταυτόσημες οι 18 και οι 19 και αυτές οι δύο, 18 και 19. Υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν. Μετά τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Οι δύο υπέρ. Άγκρι 2 βέβαια, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Άγκρι 3, πρέπει και αυτή να την ψηφίσουμε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Και τώρα η τροπολογία 3, εντάξει, υπέρ, κατά, Έλεγχος. Ψηφίζουμε την τροπολογία 3 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας λοιπόν. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 47 υπέρ, 9 εναντίον, 2 αποχές. Και περνάμε στη δεύτερη τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία πάλι. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Λείπουν κάποιοι που δεν συμμετείχαν. Προφανώς συμμετέχουν όλοι στην ψηφοφορία. Τέρμα ψηφοφορίας λοιπόν. Αποτέλεσμα 41 υπέρ, 9 εναντίον, 4 άποχες. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, στον κύριο Αντρέ Περέγιο Ροντρίγκεθ. Θερμά συγχαρητήρια κύριε Ροντρίγκεθ για τους πολλούς αυτούς, πολλούς ε, φρουτοχυμούς, ε, τους αυθεντικούς και τους άλλους που μπορεί να αγοράσει κανείς ε, στην αγορά. So, again... Λοιπόν, περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία για το υπαριθμό 10, παρακαλώ. Esther de Lange, παρακαλώ. Δεν συμφωνώ πάντα με τον Κασλίτερ, αλλά όταν έχει δίκιο, έχει δίκιο. Κάναμε αυτή την ψηφοφορία, πρέπει να θέσουμε το ζήτημα στην νομική υπηρεσία, γιατί ε, έτσι πρέπει. Είναι σχετικό ε, μόλι ψηφίσαμε να, κάτι το να επιτρέψουμε κάτι το οποίο έχει ήδη απογορευτεί δηλαδή η προσθήκη ζάχαρη σε φυσικό χυμό. Είναι σαν να λέμε ότι δεν υπάρχει φάρμακο σε αυτό το νερό, προφανώ γιατί απαγορεύεται. Αλλά εμεί έχουμε αντιστρέψει τη λογική. Λέμε ότι θα, ε, θα έχουμε ε, θα έχουμε μια προσθήκη επιγραφής ε, για την ή προσθήκη ζάχαρης, αλλά όχι για τη λακτόζη. Και αυτό είτε πρόκειται για προσθήκη ζάχαρης, είτε για χυμό ε, Και με προς... Ε, με εκπλήσουν ε, οι σοσιαλιστές συνάδελφοι που πάντα θέλουν να υπάρχει διαφάνεια για τον ε, καταναλωτή, αλλά τώρα δεν, δεν τους νοιάζει. Το ξέρω, Δάγμα, ότι ε, σας ενδιαφέρει. Αλλά αυτό το ερώτημα του Κάρου Λίτρης α το θέσουμε στην νομική υπηρεσία. Είναι λογικό αυτό που κάνουμε. Αλλά και προ την Επιτροπή ευθυγραμμίζεται με την αντίστοιχη οδηγία. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε για αυτό το σχόλιο, Εστέρ. Αύριο από πλευρά σα συντονιστή θα μπορέσει αυτό να αποσαφινιστεί και σε σχέση και με την νομική υπηρεσία. Κάπω, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα πράγματα πρέπει να αποσαφινιστούν, να έχουν αποσαφινιστεί πιο πριν. Αύριο το πρωί θα το δούμε. Α προχωρήσουμε με την ψηφοφορία τώρα για το θέμα 10 οι μεταδιδόμενες σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες, μεταδιδόμενες σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες, μη σι έψιλον. Η συγγήτρια η Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ για αυτό το θέμα. Περνάμε στην ψηφοφορία λοιπόν γι' αυτό. Παγιωμένη ολοκληρωμένη τροπολογία μόνο ένα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίθηκε. Ολοκληρωμένη Consolidated 2 υπέρ κατά αποχές και αυτή εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στις, ε, στα επιμέρους εδάφια, στις παραγράφους. Αρχικό κείμενο πρώτα, με προφορική τροποποίηση για την παράγραφο 4 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 7, υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές και αυτή απορρίφθηκε εντάξει να ελέγξουμε ωραία 8 ψηφίζουμε και άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Απορρίφθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίφθηκε. Πάμε στην τροπολογία 11. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Τροπολογία 10. Με προφορική τροποποίηση. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίθηκε. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 13 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Ε, κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 16 υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε. 21 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε. 22 υπέρ κατά άποχες έλεγχος. Ψηφίζουμε την 22. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας λοιπόν. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 29 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 32 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 30 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 31 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 33 και 34 ταυτόσημες υπέρ αυτών κατά άποχες απορρίφθηκαν 35 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε 36 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε Αιτιολογικές σκέψεις, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε, 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε, αρχικό κείμενο, με προφορική τροποποίηση, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε, η τρία τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε, τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Και τώρα φτάσαμε στην τελική ψηφοφορία που άρχεται η ψηφοφορία τώρα ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 56 υπέρ, κανείς εναντίον, μία αποχή. Συγχαρητήρια στην κυρία Ροτ Μπέρεντ για τις μεταδιδόμενες σπογκώδεις εγκεφαλοπάθειες, μισή έψιλον. Ε. Πώς είπατε? Πρόεδρε, παρακαλώ όλοι μας την τροπολογία 22 της κυρίας Αντωνέσκου που εγκρίθηκε σήμερα εδώ με μεγάλη πλειοψηφία από πλευράς ε, της Ευρωβουλής που την έρευνα για post-mortem μεταθανάτιες αυτοψίες ζητεί ζητώ να το ξαναδούμε για την Ολομέλεια. Καλύτερο θα ήταν να μην γελιοποιηθούμε έναντι των πολιτών μας, διότι Αυτά τα, αυτές οι δοκιμές post-mortem, αυτές ε, οι εξετάσεις γίνονται εδώ και 12 χρόνια. Με ξεχωριστή ψηφοφορία στην Ολομέλεια να διαγράψουμε αυτό το σημείο. Εντάξει, ευχαριστώ. Αυτή την πληροφορία θα την διανύμει και θα την διαδώσει η, ε, η συγγήτρια μέχρι την Ολομέλεια να το ξανασκεφτούμε όλοι αυτό. Πολύ καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη και περνάμε τώρα στην παγκόσμια καταπολέμηση της παράνομης αλληλείας και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η η κυρία Άννα Ροσμπαχα και που συνέταξε αυτή την έκθεση από πλευρά Επιτροπής Αλίας. Περνάμε τώρα στην ψήφιση. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 2. Εγκρίθηκε. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 7 σε τμήματα ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Η τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 11 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 12 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε 13 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε 14 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε 15 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 21 καταπίπτει, 22 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Η καταπίπτει, 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε, 26 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίθηκε. Το έχει ήταν υπέρ, έτσι. Εγκρίθηκε λοιπόν. Πολύ ωραία. Πάμε στην τελική ψηφοφορία τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας λοιπόν. Αποτέλεσμα 52 υπέρ. Κανείς εναντίον καμία αποχή. Θερμά συγχαρητήρια κυρία Άννα Ρόσμπαχ. Τα ψάρια θα χαρούν ιδιαίτερα σήμερα μετά από αυτήν την ψηφοφορία. Ευχαριστούμε και τη Γραμματεία και τους χειώδεις εισηγητές. Μετά έχουμε την επόμενη ψηφοφορία. Κινητικότητα και ένταξη ατόμων με αναπηρίες, με ειδικές ανάγκες. Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες μέχρι το 2020. Η ο κύριο Ορέστε Ρώση. Μάλιστα. Τι έχουμε εδώ. Έχουμε μία ολοκληρωμένη consolidated τροπολογία, την υπαριθμόν 6. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Μετά πάμε στην τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 16. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 12 και 14 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Μετά έχουμε συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ολοκληρωμένη τροπολογία 3 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 34 σε τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 36 υπέρ κατά αποχές και αυτή εγκρίθηκε. Ταυτόσιμες 38 και 23 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμφιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 41 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ολοκληρωμένη τροπολογία 5, consolidated 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 50 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε. Η 51 υπέρ κατά άποχες έλεγχος. Ψηφίζουμε την 51, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πάμε στην τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 2 υπέρ κατά αποχές και αυτή εγκρίθηκε και έτσι Φτάσαμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορία. 49 υπέρ, κανείς εναντίον, μία αποχή. Θερμά συγχαρητήρια στον Ορέστε Ρώση για αυτή την έκθεση. Θερμά συγχαρητήρια. Το 13 ήδη το έχουμε διευθετήσει με ψηφοφορία. Πάμε στο 14. Προφορική ερώτηση είναι αυτό για τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά <clears throat> τις ρυπογόνες και μη βιώσιμες πρακτικές. Εδώ έχουμε την ψήφιση. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της προφορικής ερώτησης λοιπόν κατά της προφορικής ερώτησης. Πρέπει ηλεκτρονικά να ελέγξουμε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά γι' αυτό. Άρχεται η ψηφοφορία. Ναι, πολύ αργά. Λοιπόν, και πάλι ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Όλο και λιγότεροι γίνονται. Τέλος ψηφοφορία. 26 υπέρ, 20 εναντίον. Η προφορική ερώτηση λοιπόν υπερψηφίστηκε και θα κατατεθεί. Και Κορίν Λεπάζ μπράντι μάλιστα. Διευθετείτε αυτό έτσι. Περνάμε λοιπόν τώρα στο 15 της ημερήσιας διάταξης. Συνολική προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών των βλαπτικών αερίων εκτός από το διοξίδιο του άνθρακα. Θα πρέπει να ψηφίσουμε και γι' αυτό, για αυτή την προφορική ερώτηση δηλαδή. Ποιοι είναι υπέρ του να κατατεθεί αυτή η προφορική ερώτηση. Κατά. Αποχές. Με μία ψήφα εναντίον και μία αποχή εγκρίθηκε. Έχουμε και το σημείο 16 τώρα. Μία αποτελεσματική στρατηγική για τις πρώτες ύλες στην Ευρώπη. Έχουμε δύο ψηφοφορίε για το 15. Την προφορική ερώτηση που εγκρίναμε πιο πριν και τώρα πρέπει και πάλι να διευθετήσουμε κάτι για τη συζήτηση να ψηφίσουμε που προτίθενται να διεξαχθεί οι ετούντες. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο προς τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος κατανοεί και λέει για τη συζήτηση για το σχέδιο ψηφίσματος. Συζήτηση που θα διεξαχθεί. Εντάξει. Οι συντάκτε θα έπρεπε να ζητήσουν τον λόγο να παρεύουν πρώτοι και να κάνουν την εισαγωγή για αυτό το ψήφισμα. Ποιο θα κάνει την εισαγωγή λοιπόν τώρα. Ο κύριο Κυλακάκης. Παρακαλώ έχετε τον λόγο κύριε Κυλακάκη. Well, thank you, Mr. President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για ένα σημαντικότατο ψήφισμα. Μέσω της δικής σας πρωτοβουλίας καταρχάς διαπιστώσαμε ότι τα καυσαέρια που προέρχονται από ε, άλλου τύπου εκτός από το διοξίδιο του άνθρακα διακόπτει ο κ. Παρακαλώ λίγη ησυχία για να ακούσετε τον εισηγητή. Ε, είπαν όνομα. Να επανέλθω λοιπόν στο θέμα μας. Είδαμε ότι αέρια εκτός του διοξιδίου του άνθρακα μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Είδαμε επίσης ότι και οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι παγκόσμιες πρωτοβουλίες για αυτά τα αέρια δεν χαρακτηρίζονται από πάρα πολύ προσπάθεια και ουσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είδαμε με το HFC 23, αλλά διακόπτει πάλι ο κύριος Κυλακάκης. Αν συνεχίσει ο κόσμος να ομιλεί δεν υπάρχει κανένας λόγος για μένα να συνεχίσω. Παρακαλώ για μια ακόμη φορά λίγη ησυχία. Έχει σημασία το θέμα από όσο μπορεί κανείς να πιστεύει, να θεωρεί. Μπορούμε να πετύχουμε θετικά πράγματα στον τομέα των κλιματολογικών αλλαγών. Έχουμε σοβαρότατα προβλήματα και παγκόσμια και στην Ευρώπη και θα πρέπει να παρέμβουμε και στον τομέα των HFC όπως επίσης και άλλων καυσαερίων μη προερχομένων από τον άνθρακα. Το ψήφισμα συνεπώς αυτό και αυτή η προφορική ερώτηση έχουν σαν στόχο να προκαλέσουν την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο τι θα πρέπει να γίνει και να πιέσουν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσεις για πιο ισχυρές πολιτικές και μέσω του πρωτοκόλλου του Μοντρέ και εδώ στην Ευρώπη. Έχουμε μιλήσει για το Ευρωπαϊκό ETS. Είδαμε ποιες είναι οι δυσκολίες, είδαμε ποια είναι τα λάθη που έχουν γίνει στο εσωτερικό του ETS. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο τομέα εκτός του ETS, όπου μπορούμε να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα για το κλίμα, και ίσως εμείς να μειώσουμε και το τίμημα το οποίο καλούνται να πληρώσουν οι βιομηχανίες για την επίτευξη των στόχων που έχουμε. Το θέμα λοιπόν είναι σημαντικότατο και ελπίζω το σύνολο της Επιτροπής μας να υποστηρίξει την πρωτοβουλία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα ήθελε το λόγο. Ο Chris Ντέιβις. Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ε, αυτή την παρουσίαση του κυρίου Σκυλακάκη. Συμφωνώ απόλυτα με ό,τι έχει υποθεί και εμεί εστιάζουμε, στο, εστιάζουμε στο διοξείδιο του άνθρακα και ε, ξεχνούμε ότι άλλα προϊόντα είναι πολύ χειρότερα. Από πολλά άλλα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στην ε, κοινωνία μας σήμερα. Είναι σημαντικό λοιπόν να το κοιτάξουμε από διαφορετική οπτική γωνία ε, και έτσι να συμπεριλάβουμε στο πεδίο προσοχή μα και, άλλα, και άλλους ρήπους. Ευχαριστώ κύριο Πρόντι. <clears throat> Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ πλήρως με την πρόταση. Συμφωνώ λοιπόν και θα ήθελα να πάμε λίγο περισσότερο, λίγο παραπέρα. Να πούμε ότι και κάποιοι τομείς ε, της οικογένειας των γενετικά τροποποιημένων θα μπορούσαν να είναι πολύ σημαντικά μέσα για την ανείχνευση αυτών των αερίων στην ατμόσφαιρα μέσω της ικανότητάς τους να μας δώσουν μια χωρική διάρθρωση των συγκεντρώσεων αυτών των αερίων η οποία θα μπορούσε να είναι σημαντικότατη για να ανοιχνεύσουμε τις πηγές, ιδιαίτερα τις πολύ συγκεκριμένες και σε συνέχεια εκπέμπουσες πηγές. Λοιπόν, θα ήθελα στη συνέχεια λοιπόν να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν για την καταμέτρηση αυτών των συστατικών που είναι πάρα πολύ σημαντικά σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα οποία θα πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα πάνω στα οποία να βασίσουμε την εκστρατεία μας κατάργησης ή μείωσης αυτών των αερίων να πω εδώ συμπληρωματικά ότι υπάρχουν ορισμένες γεωργικές πρακτικές σχετικά με, που έχουν σχέση με το άζωτο και τα οποία θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη σχετικά με τα αποτελέσματα τα αρνητικά που έχουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου αυτά τα αέρια. Άντε. θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου γιατί τα μέλη της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής δεν, είχαν, δεν έχουν ακόμα εκφράσει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν έχουν αντιδράσει σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και με αυτές τις πρωτοβουλίες. Νομίζω λοιπόν ότι ο κύριος συνάδελφος, ο εισηγητής, πράγματι προσπαθεί, αν θέλετε, σε ένα κλίμα αδιαφορίας να προχωρήσει το θέμα του, γιατί πρόκειται για αέρια τα οποία εν πωλής ίσως είναι και πιο επιθετικά και πιο τοξικά από ότι το διοξίδιο του άνθρακα. θεωρείται σε ορισμένου τομείς 12.000 ε, πιο, επικίνδυνα, πιο αυτά τα αέρια από ότι το διοξίδιο του άνθρακα. Εν πάση περιπτώσει με ένα σύστημα φορολογικό ε, δεν, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε μεσοπρόθεσμα ε, να καταπολεμήσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Πάντως το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Έχουμε περιορισμένα μέσα στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσαμε το θέμα μέχρι τώρα δεν ήταν σε καμία περίπτωση ικανοποιητικός έχουμε μιλήσει για τα ποσοστά μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, έχουμε ασχοληθεί εν πάση περιπτώσει σχεδόν αποκλειστικά με το διοξίδιο του άνθρακα, ενώ υπάρχουν και άλλα καυσαέρια τα οποία είναι σαφές ότι θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και θα πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να τροποποιήσει επιτέλους ένα σύστημα το οποίο δυσλειτουργεί. Ελπίζω λοιπόν να αντιμετωπιστεί σε κάποια φάση το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με την πρόταση ψηφίσματος. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε περισσότερο και στα υπόλοιπα αέρια του θερμοκηπίου. Βεβαίω, αυτό δεν πρέπει να έρχεται σε βάρος ε, των φιλοδεξιών μας για την μείωση των επιπέδων διοξιδίου του άνθρακα. Αλλά πρέπει να ε, επιστήσουμε την απαραίτητη προσοχή και στα υπόλοιπα αρέτη θερμοκηπή. Πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι, μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την πρόταση, να μην ε, επιμείνουμε προβολικά στο διοξίδιο του άνθρακα, μπορούμε να μιλούμε και για άλλα ε, αέρια όπως το μεθάνιο που είναι 24 φορές ε, πιο ισχυρό με 24 φορές πιο δυσμενείς επιπτώσεις σε σχέση με το διοξίδιο του άνθρακα. Και έτσι είναι σημαντικό εδώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Μπέτετ Χαλμεσφάχτ αρχικά και μετά ο Ντρέ Ζουμπέρ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή συμμερίζεται τι ε, ανησυχίε ε, για τα υπόλοιπα αέρα του εκτό από το διεξοδιο του άνθρακα. Αυτό είναι ξεκάθαρο και από τον οδικό χάρτη για την ε, ε, οικονομία χαμηλού άνθρακα μέχρι το 2050. Εκεί αναφέρεται ότι τα υπόλοιπα αέρα του θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθούν από το κατά 70 έως 78% το 2050 σε σχέση με τα επίπεδα 1990. Επομένω, συμφωνούμε και εμεί λοιπόν ε, ε, με όσα υπόθηκαν για τα υπόλοιπα του οποίου εκτό από τα του άνθρακα. Θα ήθελα επίση να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη υιοθετήσει ορισμένε πολιτικέ, όπω ο κανονισμό ε, για τα υπόλοιπα, ε, για άλλα αέρια ή για τους ε, υδροφθοράνθρακες ε, στον κλιματισμό. Υπάρχει λοιπόν ήδη ισχύουσα νομοθεσία που ήδη μειώνει σημαντικά τις ε, υπόλοιπες αυτές εκπομπές. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω δράση. Από το 2009 η Επιτροπή έχει ε, εκφράσει ανοιχτά ότι είναι σημαντικό να ε, περιορίσουμε την αυξανόμενη χρήση των ε, HCFCs αλλά και διαπραγματεύθηκε υπό το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ άλλες προτάσεις για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για να περιορίσει τη χρήση των HCFCs, συμπληρώνοντας έτσι τις συμφωνίες του UNFCCC. Ταυτόχρονα, αναθεωρούμε αυτή τη στιγμή τον κανονισμό ε, για τα fluorinated ε, αυτά αέρια και εξετάζουμε διαφορετικές ε, επιλογές για περαιτέρω μελλοντικές ενέργειες που συμπεριλαμβάνει και την πιθανότητα μείωση των HCFCs στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι ένα από τα σενάρια τα οποία εξετάζει η Επιτροπή. Υπάρχει λοιπόν πρόοδο. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Euh, Ευχαριστώ, συνάδελφό σας. Κύριε ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να δώσω ορισμένες ε, περαιτέρω πληροφορίες για το τροποσφαιρικό όζον και την μαύρη εθάλη που ήδη πάγεται επίσης στο πεδίο των ενδιαφέροντων με εδώ. Δύο πληροφορίες θα ήθελα να σας δώσω για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις υπό την αντίστοιχη σύμβαση. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκάθαρα διαπραγματεύεται ε, κείμενο που αφορά την Εθάλη. Δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση, όμως ε, υπάρχουν σενάρια για την ε, ανάληψη με για τη μείωση των εκπομπών εθάλης σχετικής στρατηγικής αλλά και αξιολόγηση των επιπέδων εθάλη ε, στι ε, στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι διαπραγματεύσει ε, θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2011 και ενδεχομένως να καταλήξουν σε ένα τροποποιημένο πρωτόκολλο το οποίο θα τεθεί σε ισχύ σε μερικά χρόνια. Έθελα λοιπόν να πω ότι η Επιτροπή ηγείται αυτών των διαπραγματεύσεων εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένονται ορισμένα αποτελέσματα μέχρι τα τέλη του χρόνου. Δεν έχουν όμως ληφθεί ακόμα αποφάσεις. Περαιτέρω, η Επιτροπή έχει αποφασίσει να αναθεωρήσει την θεματική στρατηγική ε, του για το 2005 και να επιστρέψει μέχρι το 2013 το αργότερο που θα συμπεριλαμβάνει ε, και συγκεκριμένα στοιχεία και εκεί θα εξετάσουμε και την εθάλη. Υπάρχουν αρκετέ λοιπόν διαδικασίες που συνεχίζονται, ε, των οποίων ηγείται η Επιτροπή που μπορούν να επηρεάσουν τις μελλοντικέ μας πολιτικές ε, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σκυλακάκη. Yes, I would like to θα ήθελα να πω ότι κατά την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού, Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Οργανισμού πολύ ε, πολύ πρόσφατα, στις 12 Μαΐου έγινε αυτό, αναφέρεται ότι ε, ο κανονισμός ε, των φθοριούχων αερίων όπως έχει ως τώρα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις ε, συγκεκριμένα ε, λόγω της ε, χαμηλής συμμόρφωσης δραματικά χαμηλής συμμόρφωσης με τις διατάξεις αυτές. Θα ήθελα απάντηση από την Επιτροπή. Ο κύριος Πρόντι. Environmental Investigation Agency, not Europe. Environmental Investigation Agency, λοιπόν. Rifarmi al secondo intervento della να αναφερθώ σε αυτά που είπε η δεύτερη, ο δεύτερος ομιλητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ε, επιρροές στον τομέα της υγείας και στον τομέα του κλίματος για την εφάλη η οποία βρίσκεται ε, στην ατμόσφαιρα. Είναι απαραίτητο να δούμε ποιες είναι οι πηγές και να δράσουμε στον τομέα των ε, πηγών. εκεί όπου υπάρχουν ε, και αναφέρομαι σε ε, σωματίδια κάτω των δύο μικρομέτρων. Γιατί εκεί ακριβώς δημιουργούνται προβλήματα στις ε, κυψέλες των πνευμόνων από τα συγκεκριμένα σωματίδια. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την εκπομπή αυτών των σωματιδίων στην πηγή τους γιατί επηρεάζουν αρνητικά την υγεία, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα σύνολο μέτρων τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Υπάρχουν ακόμα δυστυχώς πηγές ιδιαίτερα βλαβερές από τη μία στις ε, αστικές περιοχές όπως από τις ε, δίχρονες μηχανές με την ε, μερική ανθρακοποίηση του ε, ελαίου το οποίο παραμένει στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο σωματιδίων. Και αυτά τα σωματίδια έχουν μεγάλη διάρκεια παραμονή στην ατμόσφαιρα. Επίσης υπάρχουν προβλήματα από την καύση ξυλίας που είναι μια πολύ σημαντική πηγή αυτών των σωματιδίων και παρουσιάζουν επιπτώσεις και στον τομέα της υγείας και στον τομέα των κλιματολογικών αλλαγών. Να υπογραμμίσω επίσης πως μια πηγή πάρα πολύ σημαντική αυτών των σωματιδίων είναι το λεγόμενο flaring, η απότομη καύση, ιδιαίτερα στα, στα σημεία εξόριξης πετρελαίου. που καίει το αέριο το οποίο ξεχωρίζεται από το πετρέλαιο το οποίο αντλείται. Συνεπώς λοιπόν ε, γι' αυτό το μονοξίδιο του άνθρακα βέβαια είναι πιο αποτελεσματικό από το μεθάνιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλές ποσότητες οι οποίες δυστυχώς ε, ε, εκλείονται στην ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει αντικείμενο εξέτασης γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τα μικρά σωματίδια, τα λεπτά σωματίδια, τα οποία είναι υπεύθυνα για ένα μεγάλο ε, ποσοστό των προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από τις εισπνοές. Ευχαριστώ κύριε Πρόντι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να δώσει κάποιες απαντήσεις στην ερώτηση του κύριου Σκυλακάκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αναθεώρηση του κανονισμού για τους χλωροφλοράνθρακες, τους οποίους ξεκινά τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζει τις επιπτώσεις του ισχύοντος κανονισμού και εξετάζει επίσης και κάποιες περαιτέρω επιλογές που μπορεί να γίνουν για να πετύχουμε περισσότερα. Στις προσπάθειες τις οποίες έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι σαφές ότι ο παρόν κανονισμός έχει και θα εξακολουθήσει να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη μείωση των εκπομπών. Είναι επίσης αλήθεια ότι υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη που είναι πολύ πίσω στην εφαρμογή του κανονισμού και για να επηρεάσει θετικά ο νέος κανονισμός θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες τις οποίες κάνουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει προς την κατεύθυνση αυτή. Όπως σας είπα και στην πρώτη μου παρέμβαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί για την προϊούσα χρήση των χλωροφθοράνθρακων και εξετάζει κάποιες επιλογές για μέτρα σοβαρά τα οποία θα μειώσουν τη μόλυνση από τους χλωροφθοράνθρακες και πιέζουμε και σε διεθνές επίπεδο να υπάρξει μια σφαιρική συμφωνία για την κατάργησή τους στα πλαίσια του πρωτοκόλου του Μοντρεάλ. Κύριε Σκυλακάκη, θέλετε κάτι να προσθέσετε. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 24η Μαΐου στις 7 το απόγευμα και θα ψηφίσουμε στις 15 Ιουνίου την Ολομέλεια, θα φτάσουμε τον Ιούλιο. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης σήμερα το πρωί, είναι το σημείο 16. 9 το πρωί, α, στις 7 το απόγευμα, όχι στις 9 το πρωί. Περνάμε λοιπόν τώρα στο 16, μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πρώτες ύλες. Η κυρία Μέρκης είναι η συγγήτριά μας και της δίνω το λόγο. Μέρκης. Thank you, Madam Chair. The raw materials... Ευχαριστώ. Η στρατηγική για τις ε, πρώτες πολύ σημαντική στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ξαναρχίζει όλη αυτή η υπόθεση μετά από μερικά χρόνια από την Ήτρε. Ε, πολύ ε, σημαντική πρόκληση, αυτή από πολλές ε, πτυχές. Εφόσον υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον για αυτή την ε, έκθεση. Θα ήθελα να εστιάσω ώστε να το περισσότερο στην ε, περιβαλλοντική πτυχή. Βεβαίως υπάρχουν και πολλές άλλες ε, που, στις οποίες δεν θα αναφερθώ, το γνωρίζω αυτό. Προς το παρόν ας εστιάσουμε στις περιβαλλοντικές πτυχές των πρώτων Με τις... Εγώ ακολουθώ την εξή προσέγγιση. Είναι καλό να υπάρχει εστίαση ε, στους ορυκτούς πόρους, βιωτικούς και μη βιωτικούς πόρους. Όχι μόνο λοιπόν στους ορυκτούς πόρους, αλλά και στο, ε, στο μαλλί, στην ξυλία, γιατί ορισμένες φορές ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις διαφορετικές αυτές ε, πλευρές. Όμω, όλες αυτές οι ύλε αξιοποιούνται ε, κατά το δυνατό. Κάποιες φορές όχι. Με την βιομάζα, για παράδειγμα, έχουμε όλους αυτούς τους στόχους να το χρησιμοποιήσουμε για την ενέργεια και μετά ε, αρχίζει η καύση του, ε, που δεν ε, επιφέρει απαραίτητα την πρόσθετη αξία. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για φάρμακα. Υπάρχει λοιπόν ε, μεγαλύτερη αξία από ό,τι ε, παράγεται με την καύση του. Γιατί μετά την χρήση του για την παραγωγή φαρμάκων μπορεί ακόμα να, να αξιοποιηθεί μέσω της καύσης του. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια σωστή ε, ιεράρχηση των πρώτων υλών χωρίς πάντα να θέτουμε σε κίνδυνο το περιβάλλον. Έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση αλλά και να βρούμε τον ανταγωνισμό, αν θέλετε, για διάφορες όλες, για διαφορετικές χρήσεις. Να ακολουθήσουμε την προσέγγιση του κύκλου ζωής των πρώτων υλών. Ήδη βρισκόμαστε καθοδόν με τις ε, οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό. Πρέπει όμως να συζητήσουμε και την παράταση του κύκλου ζωής ε, της ε, πρώτης ύλη και του προϊόντος θα πρέπει να υπάρχουν οικονομικά κίνητρα για την παράταση αυτού του κύκλου ζωής και να πείσουμε τους καταναλωτές ε, να ε, αγοράσουν ένα προϊόν υψηλότερης ποιότητας και έτσι να παρατείνει τον κύκλο ζωής ε, του προϊόντος και, του προϊόντος και της πρώτης Βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τις επιπτώσεις της εξόριξης, αλλά και για τι ε, δυνατότητες ανακύκλωση. Η επαναχρησιμοποίηση δεν αναφέρεται σχεδόν ποτέ. Ορισμένες φορές η επαναχρησιμοποίηση δεν είναι ο πιο ε, ενεργειακά αποδοτικός τρόπος ε, διαχείριση μια πρώτη ύλη, αλλά συνδυάζοντα τον οικολογικό σχεδιασμό και την απεναχρησιμοποίηση, Ε, μπορούμε έτσι να έχουμε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την παράταση του κύκλου ζωής ε, τη πρώτη ύλη. Και όχι μόνο να κοιτάζουμε την ανακύκλωση, αλλά και την ε, επαν, γιατί αυτό μας δίνει ακόμα περισσότερη προστιθεμένη αξία. Τώρα για την στρατηγική για τις πρώτες ύλες. Αν ε, δούμε πώς ε, χειριστήκαμε τους συνδυακούς στόχους, μπορούμε να αντλήσουμε μαθήματα από εκεί και να βρούμε στόχους αποδοτικότητας στην ε, χρήση των πρώτων υλών. Έναν στόχο του 3%. Εάν δούμε την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, βλέπουμε ότι θα πρέπει να, να αντιστρέψουμε αυτή την καμπύλη και γι' αυτό καλύτερο θα, ακόμα θα είναι να θέσουμε και ένα στόχο. Να αποσυζεύξουμε την χρήση των ε, πρώτων υλών από την οικονομική ανάπτυξη. Και ε, προς το παρόν ε, μετρούμε την χρήση των πρώτων υλών από, από την κατανάλωση, αλλά αυτό θα πρέπει να αλλάξει. μπορούμε να αντλήσουμε μαθήματα από διάφορα πρότυπα. Για παράδειγμα, το πρότυπο μίσθωση αντί ιδιοκτησία, όπου τα προϊόντα εκμισθώνονται αντί να ε, παραχωρείται η ιδιοκτησία. Ε, επίσης, να αυξήσουμε την ε, ευθύνη ε, του παραγωγού. Αν θέλουμε να προωθήσουμε την αποδοτικότητα των πρώτων υλών, θα πρέπει να ανοίξουμε αλλά και να κλείσουμε πόρτες. Σήμερα βλέπουμε ότι πολλές πρώτες και με δική μας ευθύνη εξαφανίζονται ξαφνικά σε μία χωματερή ή και σε έναν καυστήρα. Θα πρέπει όμως να κλείσουμε αυτή την πόρτα της της Και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να ανοίξουμε άλλες πόρτες, να βρούμε νέες δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης της πρώτης ύλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής ε, της ε, ε, οδηγίας για τις χωματερές. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, το συντομότερο δυνατόν να καταργηθούν αυτέ οι χωματερέ και ο στόχο είναι η επαναχρησιμοποίηση τη πρώτη ύλη. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχει έρθει η ώρα να το κάνουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δώσουμε αξία ε, στην πρώτη ύλη. Γιατί εάν απαγορεύσουμε ε, τις χωματερές, άμα δεν έχει αξία η πρώτη ύλη, τότε αυτό που θα θα είναι παράνομο. Χρειαζόμαστε περαιτέρω εξέταση λοιπόν, για να μην πάμε από τις νόμιμε χωματερές στι παράνομες χωματερές. Γι' αυτό ε, έχω προτείνει και ένα διαφορετικό οικονομικό πρότυπο. Επίσης πρότεινα να δούμε αυτό που πρότεινε ο κ. Βουτικόβα για διαφορετική φορολόγηση. μπορούμε να εξετάσουμε τις επιπτώσεις ε, φορολόγησης ε, των ορυκτών πόρων, ε, του νερού και της χρήσης γης. Στην πράξη θα δίναμε αξία στο υλικό αυτό και έτσι προωθούμε την επαναχρησιμοποίησή του. Με την ψηλία έχουμε δει ότι το FFC, αυτή η αλυσίδα, είναι πολύ αποδοτική. Τα υλικά αυτά τα χρησιμοποιούμε με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Αν αυτό ισχύει, τότε γιατί το κάνουμε και με άλλες πρώτες ύλες. έχουμε αυτά τα ε, ματωμένα διαμάδια και τους πολύτιμους λίθους, γιατί ξέρουμε ότι αυτές ε, οι, οι πρωτεσίλες προέρχονται από εγκαταστάσεις εξόριξης ε, που, που δεν τη χάνουν και τις καλύτερες διαχείρισης. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι αρκετά σημεία δεν έχω αναφερθεί σε αυτή τη γνωμοδότηση το γεγονός ότι υπάρχει, ε, υπάρχουν δυσκολίες ε, με τα, τους χώρους Natura 2000 και την εξόριξη, γιατί η εξόριξη επιτρέπεται στους χώρους Natura 2000. Στην Ευρώπη είμαστε υποχρεωμένοι να στραφούμε στους δικούς μας πόρους και στις δικές μας δυνατότητες εξόριξης βλέπουμε ότι υπάρχει η φυσική ε, τάση να στρεφόμαστε προς τις ε, άδειους χώρους, αν θέλετε, και τόπους που δεν ε, αξιοποιούνται με κάποιον άλλον τρόπο και κατά κόρον τους προστατευόμενους χώρους από το Natura 2000. Θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά αυτό το ζήτημα και ανυπομονώ να το συζητήσουμε. Βεβαίω είναι αυτονόητο ότι το εμπόριο πρέπει να είναι δίκαιο και ότι θα έχουμε όλους αυτούς τους ε, όρους και προϋποθέσεις για το δίκαιο εμπόριο ε, και σε ό,τι αφορά την εταιρική ευθύνη. Τέλος, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα με ένα φάντασμα που έχουμε ξυπνήσει εμείς ε, των νέων τεχνολογιών ε, οι καινοτόμες τεχνολογίες ε, βεβαίως και μας ε, βοηθούν σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα στις χρήσεις του αργύρου με πολλές και διαφορετικές αναλυτικές λύσεις. Πρέπει να δούμε για παράδειγμα το, η, νανοτεχνολογία ε, πώς μπορεί να μας βοηθήσει ε, με τις πρώτες ύλες στο περιβάλλον και πώς μπορούν, μπορούμε να ανακτήσουμε αυτές τις ύλες όταν έχουν αποσυντεθεί σε επίπεδο ε, τόσο μικρό. Ανυπομονώ όμω να το συζητήσουμε, θα, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ. Κύριος Λόρεντ, παρακαλώ, σας ευχαριστούμε. Ευχαρίστω και εγώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Μάρκη, ε, την συνάδελφό μα, Να την ευχαριστήσω, είναι μια καλή κίνηση αυτή. Και για τα όσα είπε, δείχνω κάθε συμπάθεια στα όσα ανέφερε. Η, η έκθεσή τη ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση, τα λέγα. Κάπω με τρομάζει με πιο, τεράστιο, με τεράστιο ενθουσιασμό σήμερα το πρωί αγωνιστήκαμε για κάποια αριθμητικά μεγέθη 20-30% και πόσο λίγο ενδιαφέρον προκαλεί το θέμα της ασφάλειας σε σχέση με τις πρώτες ύλες στην Ευρώπη, στην Επιτροπή μας για αυτό το θέμα. Όταν θέλουμε να βοηθήσουμε σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές, αυτό θα γίνει μόνο με καινοτόμες, σε μεγάλο βαθμό καινοτόμες βιομηχανίες και βιομηχανικούς κύκλους. Για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία σήμερα ήταν ε, το ότι για δεσμευτικούς στόχους ε, υπερψηφίσαμε. Και δεν είναι απλό αυτό, π.χ. και για την ομάδα μας, όμως αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση θα έλεγα. Και έτσι Πρέπει να πω ότι μπορώ να πάω τόσο μακριά και να πω ότι το ότι σπανίζουν οι πρώτες ύλε και οι κλιματικές αλλαγές βρίσκονται στο ίδιο υψηλό επίπεδο προτεραιοτήτων για μας. Διότι αν αυτές οι κλιματικές αλλαγές γίνουν αλήθεια κάποια μέρα, τότε μόνο με υψηλής τεχνολογίας ε, συσκευές ε, και με αποτελεσματικές τεχνολογίες και συσκευές πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Αλλά υπάρχουν και φλέγοντα θέματα. Για ποιες πρώτες ύλες ε, μιλάμε για αυτή, σε αυτή την έκθεση. Και άκουσα την εξαιρετική λέξη και για την βιο, την λέξη βιολογική για παράδειγμα. Έχουμε κάθε συμπάθεια για συμπαθείς γείτονες που μπορούμε να μάθουμε από αυτούς, αλλά πρέπει να πούμε ότι τι θέλουμε στο τέλος τέλος να κάνουμε. Για μέταλλα να ενδιαφερθούμε, για ορυκτά, για χαρτί, για ξύλο, για τα εδάφη, για το νερό. Σε ποιο βαθμό επικεντρωνόμαστε σε αυτά και κατά πόσο μπορούμε να τα καταφέρουμε, διότι γενικά όλα πρέπει να τα καλύψουμε και να τα εξετάσουμε. Αλλά από όλα αυτά πρέπει σε κάποια να επικεντρωθούμε κάποια θέματα. Από την άλλη πλευρά ξέρουμε ότι αυτά τα θέματα έχουν τρεις πυλώνες για παράδειγμα. Την εξωτερική διάσταση για παράδειγμα που στον, στην Επιτροπή Εξωτερικών ε, Θεμάτων ε, εξετάζουμε και στην Επιτροπή Ανάπτυξης ε, Συνεργασίας για την Ανάπτυξη. Εκεί σίγουρα πολλά πράγματα μπορούμε να συνεισφέρουμε. Γιατί αν δει κανείς τι γίνεται από τους Ευρωπαίους, Ευρωπαίους επιχειρηματίες και εταιρείε στην Αφρική και τι κάνουν, ο ένας ή άλλος με, ας το πω έτσι, ε, ορθώνουν το ανάστημα και άλλοι ενδιαφέρονται για τις υποδομές, δηλαδή πώς μπορεί να βοηθήσει κανείς αυτή τη, ε, κάποιες περιφέρειες, κάποιες χώρες και οικονομικά και ε, για την οικονομική συνεργασία στα εξωτερικά θέματα για την ανάπτυξη έχουν πολύ μεγάλη σημασία αυτά τα θέματα. Η νοοτροπία με την οποία προσεγγίζουμε αυτές τις χώρες και αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα που έχουν όσο αφορά πρώτες ύλες για παράδειγμα. Η νοοτροπία μας πρέπει σίγουρα να αλλάξει ε, ριζικά και για τον πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδοευρωπαϊκά εδώ σε σχέση με την εισηγήτρια θα πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα πιο προσεκτικά, να δούμε σοβαρά. Εμείς για τις, ε, τους φυσικούς μας πόρους στην Ευρώπη τα καταφέρνουμε ή τι πρέπει να γίνει διαφορετικά να, για τους ε, όρους για την χλωρίδα, πανίδα βλέπουμε να υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Είχα τη μεγάλη τιμή και χαρά να έχω μια εκλογική περιφέρεια που έχει 148 χιλιόμετρα βρίσκεται από τον γείτονα, τον πιο κοντινό μας γείτονα, με καλές επιδόσεις, αλλά για τη χλωρίδα και την πανίδα τελείως διαφορετικά πράγματα γίνονται σε σχέση με την δική μου περιφέρεια του Ράιν, του Κατορίνου και για ένα ορυχείο το οποίο έκλεισε πριν από 20 χρόνια επειδή εκεί υπάρχει βιότοπος ε, και υπάρχουν απαγορεύσεις θα πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά μήπως θα πρέπει πιο ε, προηγμένα να τα αντιμετωπίσουμε στρεφόμενοι προς το μέλλον με πιο για προδιαγραφές ε, να δούμε περιφερειακά και εθνικά για αυτούς τους πόρους τι μπορεί να γίνει. Το θέμα της πολιτικής ανακύκλωσης που προανέφερε η κυρία Μακής, αυτό το θέμα με απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να σας πω την λέξη ανακύκλωση. Η λέξη ο όρος ανακύκλωση δεν έχει καθοριστεί δεσμευτικά στην Ευρώπη. Δεκάδες φορές το έχω δει και το έχω αναφέρει και δεν υπάρχει ιδιαίτερη υποστήριξη να αποσαφινιστούν αυτά. Για τα απόβλητα των ηλεκτρονικών, των ηλεκτρικών συσκευών λένε, για παράδειγμα οι ε, μέχρι 16 κιλά και υπάρχει, έχουν συλλογή, συλλέγουν 16 κιλά για παράδειγμα σε σχέση με, τον, ε, με, με, τους ε, πολίτες ε, στην Αυστρία 3 κιλά. Θα πρέπει τουλάχιστον να καταλήξουμε στα 10 κιλά από τις συλλογέ αυτές, την αποκομιδή τους. Και θα πρέπει και το κράτος να εμπλακεί για να ρυθμιστούν αυτά. Σε αυτό το θέμα της ανακύκλωσης λοιπόν και της πολιτικής ανακύκλωσης πολλά πρέπει να κάνουμε. Να ρυθμίσουμε σωστά και λεπτά ε, τις διατάξεις και τους κανονισμούς ώστε οι επιχειρήσεις, οι βιομήχανοι να μπορέσουν να κατευθυνθούν εκεί όπου πολιτικά θέλουμε εμείς να καταλήξουμε. Επανάχρηση δηλαδή, ανάκτηση και επανάχρηση. Και για τις ε, χωματερές ε, που πριν από κάμποσα χρόνια είχαμε απασχοληθεί για αυτό το θέμα και αυτό είναι σημαντικό. Και εγώ είμαι σημαντικό να κλείσουν αυτές οι χωματερές αύριο αλλά αν σκεφτεί κανείς ε, με ρεαλιστικό πνεύμα τα νέα κράτη-μέλη στην Ευρώπη, για ε, στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία δεν μπορούμε να του πούμε κλείστε αύριο τις χωματερέ, όποιο το πει αυτό και το ζητήσει δεν αναγνωρίζει τα προβλήματα. Αλλά τουλάχιστον να μην προάγουμε, να μην προωθήσουμε υπερβολικά τις ε, χωματερέ. και πρέπει να προαχθούν και οι μονάδε καύση. και μάλιστα με γενναίο τρόπο, με θάρρο ώστε να παράγεται και θερμότητα που να θερμαίνει πόλεις ε, και αστικά κέντρα και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε μια κερδοφόρα δράση. Η μίσθωση, γιατί η μίσθωση έχει ήδη ξεκινήσει. Μια πολύ μεγάλη εταιρεία εξορρυκτικών ε, μηχανημάτων, η κάτω είπα, ε, δεν μπορεί να διαθέσει στην αγορά τέτοιου είδους ε, τεράστιες συσκευές. Πρέπει να έχουμε περισσότερη δυνατότητα εξαγοράς δικαιωμάτων χρήσης όσον αφορά τη μίσθωση. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δίνοντας κίνητρα για παράδειγμα. Και ο τομέας αυτός είναι σημαντικός. Όσον αφορά τις ε, αποθέσεις ε, της ε, χωματερές, υποθέτω ότι στο μέλλον θα πρέπει να κινηθούμε προς μια κοινή κατεύθυνση, αλλά θα δείτε ότι θα βρούμε μεγάλες αντιστάσεις και αντιρρήσεις. Υπάρχουν χώρες που έχουν τρύπες ας το πούμε έτσι και τις γεμίζουν με αυτόν τον τρόπο. Χωματερές. Δεν είναι πολύ κομψό αλλά το κάνουν αυτό. Και είναι χώρες που είναι ιδρύτριες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι η τελευταία προσχωρήσασες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέα κράτη-μέλη αλλά χώρες ιδρυ, ιδρυτικά μέλη. Και όταν λέμε για αυτά τα πράγματα, τι θέλουμε, να ξανανοίξουν παλιές ε, χωματερές, ε, ή μήπω θα έχουμε κάποιες καινοτόμες ιδέες και προτάσεις να μπορέσουμε να εκπονήσουμε προτάσεις ώστε να δούμε πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά με τον καλύτερο τρόπο και πώς μπορούν να κατευθυνθούν στη σωστότερη κατεύθυνση. Πρέπει να πω ότι αυτά πρέπει να προσδιοριστούν ενεργητικά, ενεργειακά κριτήρια ενεργειακής αποδόσης και αποδοτικότητας, το ότι χρειαζόμαστε ε, μια κοινή, ας το πω σε ένα κοινό πλαίσιο, σωστό. Αλλά αν θέλουμε κάποια μεγέθη, αν αυτά θα υπάρξουν, υπάρχουν τομείς όπου πολλά μπορούν να γίνουν σίγουρα. Όμως υπάρχουν άλλοι τομείς όπου το κόστος για τη μείωση είναι πραγματικά ακραίο. Είναι θέματα που πρέπει να τα συζητήσουμε οπωσδήποτε. Αλλά αυτά πρέπει να μπορέσουν να ε, εξεταστούν. Για την ιεράρχηση των πρώτων υλών, με μια πρώτη ματιά φαίνεται ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση. Αν όμως ε, δεν υπάρξει υποστήριξη, διότι δεν θέλω να είμαστε εμείς πολιτικά υπεύθυνοι για τους τόνους χάλιβα που θα ε, χρησιμοποιούνται για παράδειγμα σε ένα ασθενοφόρο σε σχέση με ε, άλλη χρήση. Διευκολύνουν τα πράγματα λέγοντας καλύτερα να γίνεται αυτό στα ε, ασθενοφόρα παρότι για παράδειγμα στα παιδικά παιχνίδια ή στους, στα McDonald's. Πρέπει όλα αυτά να τα δούμε προσεκτικά, με συνειδητά και με μια τακτοποίηση και ιεράρχηση. Για τις ιεραρχήσεις σε, στην πολιτική για το περιβάλλον στην Ευρώπη έχουμε δυστυχώς ε, κακή πείρα. Να συζητήσουμε για την ε, ε, νέα ιεράρχηση σε σχέση με τις προτάσεις αυτές με τις ιεραρχίες αυτές είμαι πιο προσεκτικός και επιφυλακτικός αλλά την αρχή αυτή για την αλλαγή νοοτροπίας και συνείδησης την προσυπογράφω ως αίτημα φόροι για τις πρώτες ύλες και τέλη για ε, μια τέτοια πρόταση είναι βρίσκει την CDU κατά. Είμαστε κατά των φόρων. Είμαστε υπέρ των κινήτρων που θέλουμε να δώσουμε. Δεν θέλουμε να τραβήξουμε, να πάρουμε λεφτά από τις τσέπες των ε, πολιτών μας, από τους φορολογούμενους. Εν πάση περιπτώσει, συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε να συνεργαστούμε ώστε στο τέλος να έχουμε μια καλύτερη έκθεση από ό,τι αυτή τη στιγμή τώρα. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το γεγονό ότι συζητούμε εδώ πέρα αυτό το θέμα μα δείχνει ότι στο ιστορικό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει διχόνοια ε, για το πώς πρέπει να χειριστούμε το ζήτημα των πρώτων υλών. Έχουμε αυτή τη στρατηγική για τι πρώτε ύλε ε, που αναφέρεται ιδιαίτερα στην διαθεσιμότητα των ε, πρώτων και έχουμε και τον οδικό χάρτη που είναι και ένα από τα κύρια σημεία της στρατηγικής Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020, που εστιάζει στην πιο αποδοτική χρήση και αξιοποίηση των πρώτων υλών. Βεβαίω θα πρέπει να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, γιατί συνδέονται. μιλάμε και για την ε, έλλειψή τους. Τώρα το εύρος του ζητήματος, πολύ μεγάλο το εύρος, από, έχει οικονομική πτυχή. Γιατί καθημερινά βλέπουμε επιχειρήσει ε, που αντιμετωπίζουν δυσκολίε λόγω τη αύξηση των τιμών των πρώτων υλών ή επιχειρήσει που θα πρέπει να αυξήσουν τι τιμέ του ε, λόγω ε, των πρώτων υλών. Γεωπολιτική πτυχή. Πριν από μερικού μήνε είδαμε και στην Κίνα για την πολιτική που εφάρμοσε για ορισμένες σπάνιες πρώτες Και βεβαίω ε, έχουμε και την εξάλληψή τους. Γιατί όταν ε, τις ε, εξοριγνύουμε τόσο εντατικά, βεβαίως και κάποια στιγμή θα εξαλειφθούν. Αυτό είναι το εύρος λοιπόν του ζητήματος. λυπούμε που η Επιτροπή δεν αντιμετώπισε με το ίδιο ανοιχτό πνεύμα το ζήτημα αυτό, αλλά πρώτα ε, εστίασε στην διαθεσιμότητά τους. Τώρα, για μένα, εξετάζοντας την ανακοίνωση, κοιτάμε την εξασφάλιση το, της εισαγωγής ε, των ε, πρώτων υλών που παράγονται ε, στο εξωτερικό. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και μετά αυτό που θα έπρεπε να έχετε πάνω-πάνω είναι η πολύ πιο αποδοτική αξιοποίηση των πρώτων υλών που ήδη έχουμε. και όχι μόνο την μικρότερη χρήση των παρθένων πρώτων υλών, των νέων πρώτων ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να έχετε ακολουθήσει με διαφορετική προσέγγιση την ακριβώ αντίστροφη. Έχω ορισμένε ερωτήσει ε, τόσο προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και ω προ τον εισηγητή. Αρχικά, ποια είναι τα μέσα ή εργαλεία που έχουμε ως Ευρωπαίοι. Θεωρώ εξαιρετική ιδέα ε, να θέσουμε αυτό το στόχο ε, του 3% που αναφέρθηκε, αλλά ποιο θα είναι το μέσο που ε, θα χρησιμοποιήσουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοιο στόχο έχω δει και στο παρελθόν και δεν υπήρξαν αποτελέσματα. Κάτι που συνδέεται με αυτό, έχουμε πολύ μεγάλη ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία που ε, εστιάζει στην ε, καλύτερη αξιοποίηση και πιο αποδοτική αξιοποίηση κυρίως των αποβλήτων. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Άλλες χώρες απλώς πετούν το 80-90% των παραγόμενων προϊόντων ενώ άλλες χώρες δεν αναποθέτουν σχεδόν τίποτα. Όμως η εφαρμογή όλων αυτών των διαφόρων ε, ε, οδηγιών δεν είναι η βέλτιστη. Αν κοιτάξουμε την πιο αποδοτική ε, αξιοποίηση των πρώτων υλών, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάξουμε την ισχύουσα νομοθεσία και πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους στο ζήτημα της ανακύκλωσης και τα λοιπά, πώς θα βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας σε αυτό τον τομέα. Τέλος, Πρόεδρε, Ε, πολύ χαίρομαι που τονίστηκε η σημασία της βιοπικιλότητας, γιατί πολλές φορές ξεχνούμε σε αυτό το διάλογο ότι οι πιο σημαντικές ε, πρώτες ύλε ε, συνδέονται με την βιοπικιλότητα, είτε στον αέρα, στο νερό, στην ξυλία. Και έτσι θα πρέπει να έχει ε, προεξέχουσα θέση στην στρατηγική για τις πρώτες ύλε. Κλείνοντας, η πρόταση ε, σε φόρου επί των πρώτων υλών ε, θα μπορούσε να μας ενδιαφέρει, αλλά εξετάζοντας την εξέλιξη ε, των τιμών των πρώτων υλών, διαρωτώ αν θα ε, επηρέαζε θετικά την όλη υπόθεση ή αν θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις και για τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά και για άλλες επιχειρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω την Επιτροπή να, να βρει θετικά κίνητρα για να επιταχυνθεί η εκ νέου χρήση των ήδη χρησιμοποιημένων πρώτων υλών. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Σλίτερ. Ah, ah, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ την κυρία Μέρκης για μια εξαιρετική έκθεση. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό και όπως είπε ο κύριος Φλόρενς, εκπλήσωμαι κι εγώ γιατί δεν είμαστε πολύ εδώ. Εγώ έτσι κι αλλιώς όμως βρίσκομαι εδώ ακριβώς λόγω αυτού του θέματος. Όταν συζητάμε για τις κλιματολογικές συνέπειες και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα δεν συζητάμε συχνά ε, τους πόρους, τους σπάνιους τους οποίους έχουμε πλέον στη διάθεσή μας και τις πρώτες ύλες, αλλά όπως είπε και ο κ. Σχεμπράντη, θα πρέπει να μιλήσουμε γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και την αποτελεσματικότητα με την οποία χρησιμοποιούμε τα μέσα και τις ύλες τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας και αναφέρουμε εδώ και στη χρήση των γεών κτλ. Υπάρχουν τρία θέματα τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν και αυτό θα πρέπει να γίνει σε τη σωστή σειρά. Πρώτον, αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε αν η εξόριξη στο εσωτερικό της Ένωσης είναι εφικτή. Και τρίτον, να δούμε ποιος είναι ο αηφόρος και σωστός τρόπος για την αντιμετώπιση ε, ε, των προβλημάτων των πρώτων υλών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας για την ομοδότηση της κυρίας Μέρκης. Ξεκάθαρα λέει ότι απαιτούνται ε, σαφέστεροι στόχοι, αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα την αύξηση κατά 3%. Το ερώτημα είναι μιλάμε για έναν απόλυτο στόχο ή ένα σχετικό στόχο. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να είμαι απόλυτο στόχο γιατί σε επίπεδο σχετικών στόχων όχι μόνο είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς, αλλά αν έχει κανείς μια ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, την οποία δεν έχουμε τώρα, τότε υπάρχουν μειώσεις λιγότερες από ότι στις οικονομίες μας έτσι όπως λειτουργούν σήμερα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τους στόχους. Να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για απόλυτους στόχους. Ένα από τα άλλα θέματα που υπογραμμίζουν τη σημασία που έχει το θέμα είναι να δηλώσουμε ότι στοχεύουμε σε δεσμευτικούς στόχους. Όπως είδαμε και εδώ και κάποιες δεκαετίες για τις κλιματολογικές αλλαγές, ξεκινήσαμε χαλαρά και με μακροπρόθεσμα μέτρα, αλλά χρειάστηκαν συγκεκριμένα άμεσα μέτρα για να διαφοροποιηθεί η κατάσταση και τώρα το πετυχαίνουμε σιγά σιγά σε επίπεδο κλιματολογικών αλλαγών, αλλά στον τομέα της βιοπικιλότητας είμαστε σε επίπεδο στόχων για το 2020 και εδώ έχουμε τον κίνδυνο ε, να μην κάνουμε τίποτα. Όλοι λένε τι σημαντικό είναι το θέμα, αλλά όταν πρόκειται να πάρουμε συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις δεν υπάρχει καμία πρόταση. Μία από τις προτάσεις που κάνουμε λοιπόν είναι οι στόχοι για τις πρώτες ύλες να είναι τμήμα του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να βλέπουμε το πού βρίσκονται και κατά πόσο είναι υπόλογες οι χώρες, όχι μόνο στον τομέα του κλίματος αλλά και των πρώτων υλών. Πολύ σωστά αναφερθήκατε ε, και στην συγκεκριμένη οδηγία. Πράγματι εμείς θέλουμε αυτό το eco να έχει ευρύτερη εμβέλεια, γιατί ό,τι ε, προωθεί ε, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα είμαστε υπέρ για τα απόβλητα και την οδηγία πλαίσιο. Θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς εδώ. Εδώ απαιτείται να ιεραρχήσουμε το θέμα των αποβλήτων έτσι όλες τις πολιτικές στην Ένωση να αναγνωρίζουν την ιεράρχηση αυτή. Νομίζω ότι αυτό είναι ίσως και λίγο πιο σημαντικό από ότι η απλή απαγόρευση των, της εναπόθεσης αποβλήτων. Θα πρέπει να δούμε αν μια τέτοια πλήρης απαγόρευση είναι χρήσιμη γιατί μπορεί να υπάρχουν ε, και χωματερές παράνομες. Αν απαγορεύσει κανείς τις χωματερές, τότε σε αυτή την περίπτωση θα επιλέξουμε τη δεύτερη ε, πιο εύκολη λύση που είναι η καύση. Και η καύση δεν είναι και ιδιαίτερα καλή όταν μιλάμε για τις πρώτες ύλες. Συνεπώς θα πρέπει να ιεραρχήσουμε σωστά τα πράγματα γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε ε, κάποιες λύσεις, λύσεις όχι μόνο στην εναπόθεση των αποβλήτων αλλά και στην καύση που είναι προβληματικές. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε λίγο την ιεράρχηση αυτή. Τέλος για τη φορολογία. Όταν μιλάμε για φορολογία ξέρω ότι όλοι ξαφνικά γίνονται πολύ διστακτικοί για το αν είναι σωστή ή όχι μια τέτοια κατάσταση. Όταν μιλάμε όμως για την σωστή χρήση των πρώτων υλών και για τις πρώτες ύλες, η φορολογία είναι ένας από τους τρόπους που θα μας βοηθήσουν να καταστήσουμε την ανακύκλωση πιο συμφέρουσα σε σχέση με άλλες επιλογές. Η φορολογία είναι μία από τις βασικές αρχές όπου τίθεται από τη μία το θέμα των κινήτρων των τιμών και από την άλλη όλες οι πολιτικές, όλα τα πολιτικά κόμματα υποστηρίζουν ότι η φορολογία θα πρέπει να απεμπλακεί από το θέμα των θέσεων απασχόλησης και των πρώτων υλών. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή λοιπόν τώρα. Δεν ζητάμε επιπλέον φόρος, δεν ζητάμε επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις, αλλά κάποιες μετακινήσεις ε, των φόρων από την εργασία στους φυσικούς πόρους. Και εκεί λοιπόν οι φόροι μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο και πρέπει να είμαστε πιο σαφείς και ελπίζω οι πολιτικές ομάδες να συμφωνήσουν. Γιατί όταν μιλάμε για τη φορολογία καλό θα είναι να κάνουμε αυτά τα οποία λέμε και να μην μένουμε στα λόγια. Θα σας βοηθήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τους, το λόγο τώρα στους ε, μη όχι πάνω από δυόμιση λεπτά, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Υπνά. Σας ευχαριστώ πολύ. Η στρατηγική σε σχέση με τις πρώτες ύλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι φυσικές πρώτες ύλες ε, σχεδόν ε, θα εξαντληθούν, εξαντλούνται. Πρέπει λοιπόν να βιαστούμε, να ακολουθήσουμε μία πορεία για να διαμορφώσουμε τις σωστές πολιτικές η εκμετάλλευση αυτής, ε, αυτής πτυχής των πρώτων υλών δεν πρέπει να είναι ληστρική, αλλά πρέπει να συνεισφέρουμε ώστε πιο εξορθολογισμένα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πρώτες ύλες. Για αυτή την έκθεση θεωρώ ότι εδώ πολλά στοιχεία εμπεριέχονται που όλοι θα, θα τα υποστηρίξουμε. Όμως θα ήθελα να επικεντρωθώ και να αναφερθώ στα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε. Πολλές φορές αυτά τα προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί τα θεωρούμε απόβλητα. Στην ορολογία μας ε, θα ήθελα να λέμε απόβλητα είναι εκείνα τα οποία δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την παραγωγή άλλων αγαθών ή προϊόντων. Αν έτσι συμφωνήσουμε και έτσι το εννοούμε, ότι κάποιο χρησιμοποιημένο προϊόν, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έστω και εν, μέρο, εν μέρη για κάποια χρήση και ένα τμήμα αυτών των υλικών του θα μπορούσε έτσι να χρησιμοποιηθεί, θα είχαμε δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και μιας, πιο, ε, μιας ευρύτερης ανακύκλωσης. Και το θέμα των μεγαλύτερων εγγυήσεων, ε, πιο ε, μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας. Οι εγγυήσει είναι πραγματικά πολλές φορές πολύ μικρής χρονικής διάρκειας. Ε, το χρονικό διάστημα χρήσης αυτών των συσκευών 5-6 ετών πολλές φορές, αν καταφέρναμε οι ίδιοι οι παραγωγοί, οι οποίοι θα, θα υπέκυντο σε κάποιες νομικές διατάξεις από πλευράς μας, ώστε να παρατείνουν την εγγύηση για τα προϊόντα τους, ή και διαφορετικά θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Κατά την επιστροφή κάποιων ε, συσκευών μετά από πέντε χρόνια, όπως ε, και για ε, τα οχήματα, για τα αυτοκίνητα, μπορούν να επιστραφούν δηλαδή, παρότι θα μπορούσαν να, χρησιμοποιήσουν, να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω, αυτό θα ήταν μια δυνατότητα. Κάνουμε λόγο δηλαδή εδώ φυσικά για τις φυσικές πρώτες ύλες που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να μην επιβαρύνεται περαιτέρω το περιβάλλον και να μην βλάπτεται. Είναι ασύλληπτο, είναι αδιανόητο σήμερα το ότι το κόστος για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης παραγωγής για συγκεκριμένων προϊόντων βιομηχανικών κύκλων υφίσταται το περιβάλλον ζημιές που πραγματικά είναι απειλητικές για όλους μας και πλήττουν όλους. Γι' αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε με καλύτερο τρόπο ώστε η πολιτική να εστιάζεται στην ε, χρήση των πρώτων υλών χωρίς να υπάρχει επιδείνωση στους όρους ε, του περιβάλλοντος ε, όσον αφορά το ίδιο το περιβάλλον ώστε να να κληροδοτήσουμε το περιβάλλον σε καλή κατάσταση στις επόμενες γενναίες. Πρέπει λοιπόν εδώ να ε, το δούμε αυτό με τον τρόπο ώστε να αλλάξει ο ορισμός των αποβλήτων. Να τροποποιήσουμε τον ορισμό των αποβλήτων και κάθε προϊόν να μπορεί να χρησιμοποιείται ή να εννοείται ως πηγή πρώτων υλών για την ανάκτηση. Ευχαριστώ. Κύριος Πρόντι παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε σε βάθος το θέμα. Εν πάση περιπτώσει έχουμε εδώ ένα θέμα το οποίο αφορά την αηφορία γενικότερα. Άμεσα όμως. Η αηφορία θυμίζω ότι είναι στο κέντρο των αλλαγών στις οποίες εμείς θα πρέπει να προβούμε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα δίκαιο, το δίκαιο στην πρόσβαση στους φυσικούς πόρους και από την παρούσα γενεά αλλά και από τις ε, μελλοντικές γενναίες το δίκαιο αυτό θα πρέπει να ισχύει. Αυτό ακριβώς είναι και η βάση της αηφορίας. Αυτό ακριβώς είναι η ανάγκη την οποία αντιμετωπίζουμε λοιπόν. Η αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων και ταυτόχρονα μία προσπάθεια να φύγουμε από την ηλική διάσταση της κοινωνίας γιατί η κοινωνία μας βασίζεται στην χρήση του ε, ΑΕΠ που μετρά, προσμετρά την υλική παραγωγή και μόνο αυτό ε, υπολογίζουμε. Αυτή είναι μια μεγάλη αντίφαση λοιπόν την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σοβαρή αντίφαση γιατί έχουμε πλέον φτάσει στα όρια των διαθεσίμων φυσικών πόρων. Αυτός είναι λοιπόν ο βασικός μας προβληματισμός και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μια προσπάθεια να καταστήσουμε την παραγωγή μας όλο και λιγότερο υλική. Να πω ότι υπάρχουν ορισμένα υλικά επίσης τα οποία χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι αυτονόητη η διασπορά τους. Ο φόσφορος, σαν παράδειγμα, υπάρχουν υποτίθεται διαθέσιμα για 70 χρόνια, χρησιμοποιείται κυρίως σε χημικά προϊόντα όμως, τα οποία ευνοούν τη διασπορά του προϊόντος. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αλλάξει. Το ίδιο φαίνεται ότι θα γίνει και με το ασίμι. Φαίνεται ότι ε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάχυση στη χρήση και αυτό είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει αρνητικά και σε επίπεδο χημικό. Συνεπώς όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο μέλλον, μη αγνοώντας την δυνατότητα ανάκτησης των πάντων. Να δώσω ένα μικρό παράδειγμα στα χρυσορυχεία τα ποσοστά ε, εξόριξης είναι 5 γραμμάρια ανατόνο εδάφους. Στα τηλέφωνά μας εδώ, στα κινητά, έχουμε 150 ε, γραμμάρια ανατόνο συνολικά βάρος μικρών τηλεφώνων φορητών. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να αλλάξουν και θα πρέπει να τα ε, διαμορφώσουμε με διαφορετικό τρόπο, να τα προγραμματίσουμε καλύτερα γιατί από αυτά θα εξαρτηθεί η αηφορία της κοινωνίας μας στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διευρύνουμε τον ορίζοντα και σε άλλους παράγοντες, όχι μόνο στο ΑΕΠ. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό εδώ και αρκετά χρόνια. Ευχαριστώ. να συνεχίσω σε σχέση με αυτά τα οποία λέγατε για τους στόχους στον τομέα της αποτελεσματικότητας χρήσης των <clears throat> πρώτων Η έκθεσή σας είναι μια καλή έκθεση, αλλά πρέπει φυσικά να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Η παραδοσιακή λογική είναι ότι επιδιώκουμε την ανάπτυξη. Ανάπτυξη, έχουμε υπογράψει το σύμφωνο για την ανάπτυξη για να έχουμε θέσεις απασχόλησης το θέμα είναι όμως ότι η αποτελεσματικότητα χρήσης των πρώτων υλών είναι μηδενική πλέον, γιατί η Κίνα επενδύει πάρα πολλέ υποδομές και το ίδιο θα κάνει για τα επόμενα χρόνια. Και όταν μιλάμε για σφαιρική, για παγκόσμια αποτελεσματικότητα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εμείς στη Σουηδία είχαμε καλά, καλά αποτελέσματα μόνο και μόνο γιατί μεταφέραμε παραγωγές προϊόντων εκτός Σουηδίας. Και γι' αυτό καταφέραμε να έχουμε υψηλή τέτοιου είδους αποτελεσματικότητα στη χρήση των πρώτων υλών. Σε παγκόσμιο επίπεδο κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Η πρόκληση είναι μεγάλη λοιπόν. Θέλουμε να γινόμαστε σε αιτήσια βάση πιο αποτελεσματικοί. Το θέμα είναι να χρησιμοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτή για να αντισταθμίσουμε μια αναπτυσσόμενη οικονομία. Οπότε ε, τότε πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές καυσαερίων. Ακόμα και με τα σωστά μέσα για να προωθήσουμε την αποτελεσματικότητα, ποτέ δεν είναι εύκολο να αντισταθμίσει κανείς και την λογική της ανάπτυξης και τις επιπτώσεις της λογικής αυτής της θέσης απασχόλησης και στη μείωση των καυσαερίων, των εκπομπών. Είναι δύσκολο λοιπόν να έχει κανείς ε, μια αιτήσια βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατά 6% κατέτος, αν πρέπει να αντισταθμίσουμε και την οικονομική ανάπτυξη και την ε, μείωση της εκπομπής των εκπομπών. Το θέμα είναι λοιπόν αν το σύμφωνο σταθερότητας είναι ο σωστός δρόμος για το μέλλον της Ευρώπης. Ίσως για να έχει κανείς μια δίκαιη κατανομή του πλούτου θα πρέπει να προσπαθήσει να σκεφτεί τις αιτήσει αυτές βελτιώσεις και για τη μείωση του χρόνου απασχόλησης και να χρησιμοποιήσουμε το κέρδος σε επίπεδο αποτελεσματικότητας κατ' για να μειώσουμε τις εκπομπές και να επιτρέψουμε αντίστοιχες αυξήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες γιατί αλλιώς πώς θα αναπτυχθούν. Αυτό είναι το δίλημα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει μέσω της λύσης να έχουμε και θέσεις απασχόλησης και μείωση των καυσαερίων. Όλα αυτά δεν γίνονται. Και φοβάμαι ότι σαν τέτοιος ένας στόχος που θέτουμε θα μας εμποδίσει. Μακάβανε. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ και την ε, Τζουντίθ που μας, ανέφ... Ε, μας παρουσίασε μια τόσο λεπτομερή έκθεση. Δύο σημεία έχω να αναφέρω μόνο. Πρώτον, ε, στο σημείο 9... Ε, χαίρομαι που συμπεριλήφθη αυτό το σημείο εδώ, γιατί πολλές ύλες που επαναχρησιμοποιούνται προέρχονται από ορισμένες πολύ δύσκολες εντός περιοχές με απίστευτη ανθρώπινη εκμετάλλευση. Επομένω, αυτό ό,τι κάνουμε στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να καθιστά ακόμα χειρότερη τη ζωή αυτών των ανθρώπων εκεί. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, όταν εξετάζουμε το τι θα κάνουμε και πώς θα καθορίσουμε αυτή τη στρατηγική μας για τις πρώτες ύλες. Το δεύτερο σημείο αναφέρθηκαν μια και άλλοι συνάδελφοι για την συνοχή στις, ε, ε, στις ίδιες μας τις πολιτικές. Θα ήθελα να ζητήσω ορισμένε πληροφορίε από την Επιτροπή. Γιατί ε, πρόσφατα συνάντησα ορισμένου κατασκευαστέ γυαλιού ε, που είχαν συλλέξει μεγάλε ποσότητε γυαλιού για ανακύκλωση, έως ότου τοπικές αρχές στην περιφέρειά μου ε, άρχισαν να συλλέγουν ε, τα, άρχισαν την αποκομιδή των απορριμμάτων από τα πεζοδρόμια. Όμω ουσιαστικά πώ γίνεται αυτό, βάζουν το πλαστικό μαζί με το γυαλί. Και μέχρι να φτάσει το γυαλί στο σημείο τη ε, ανακύκλωση του, δεν μπορεί να ανακυκλωθεί ω γυαλί, αλλά να μετατραπεί μόνο σε μια επιφάνεια. Γιατί το, ε, το προϊόν έχει υποστεί ζημιά και βλάβη μαζί, με την κοινή αποκομιδή μαζί με το πλαστικό. Έτσι χρειαζόμαστε από την Επιτροπή να κάνει μια ανάλυση και να μας πει ποια, ποιος είναι καλύτερος τρόπος ε, για την διαχείριση της ανακύκλωσης. Αν είναι χειρότερο λοιπόν ε, οι τοπικές αρχές να στείλουν δύο διαφορετικά φορτηγά ή οχήματα για, για την αποκομιδή των ε, ε, αποβλήτων, αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε αλλά θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένε επιλογέ ε, ανάμεσα α πούμε στην περίθαλψη των ηλικιωμένων ή περισσότερη ανακύκλωση. Όμω, ε, να εστιάσουμε και σε αυτά τα ζητήματα γιατί θα, είναι πιο εύκολο να τα επιλύσουμε σχέση με άλλα. Ευχαριστώ κύριο Σάντερ. Σύντομα μπορείτε. Ε, σε ευχαριστώ πρόεδρε βρισκόμαστε σε διαφορετικά πολιτικά κόμματα, όμως παρόλα αυτά θέλω να βοηθήσω την εισηγήτρια. Με ένα παράδειγμα, πέρυσι εμείς είχαμε εγκρίνει μία πρωτοβουλία και οι σοσιαλιστές είχαν υπερψηφίσει ώστε η βασισόμενη σε κιάνιο τεχνολογία να απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μεγάλη πλειοψηφία υποστηρίχθηκε αυτή η πρωτοβουλία. Από την άλλη πλευρά, εδώ και εβδομάδες και μήνες κάνουμε συζητήσει ε, και ο Καρλ Χάιντ είχε για παράδειγμα αναφέρει το θέμα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Πώς αυτά μπορούν να συνδυαστούν και να βρεθούν σε ένα κοινό παρονόμαστη λοιπόν όταν έχουμε την συλλογή ηλεκτρικών αποβλήτων και ε, επανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση. Αν υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε αυτή τη συνιστόσα, από τον ίδιο όγκο αποβλήτων 150 φορές περισσότερο όγκο χρυσού μπορεί να κερδιθεί από ότι σε σχέση με την αναλογία σε ένα τόνο ε, γεών και ορυκτών. Μιλάμε για πολύ μεγάλη βελτίωση σε σχέση με την τεχνολογία. Από ένα τόνο ε, χώματος ή ε, γεών και ε, ορυκτών κάποια γραμμάρια κερδίζουμε 150 όμως γραμμάρια μπορούμε να κερδίσουμε από ένα τόνο ηλεκτρονικών συσκευών Πρέπει με, μεγάλη, με μεγάλο ζήλο λοιπόν να αποδηθούμε σε αυτή την προσπάθεια. Από την άλλη πλευρά, με όλα τα μέσα πρέπει οι παλαιές τεχνολογίες να απαγορευτούν. Από την άλλη όμως πλευρά, οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει να προαχθούν με κάθε δυνατότητα, με κάθε τρόπο και να προαγάγουμε και τις χρήσεις των νέων τεχνολογιών. Και σε αυτό ανήκει και η ανακύκλωση και η επανάκτηση αποβλήτων. Δύο λεπτά λοιπόν κράτησα πρόεδρε στην παρέμβασή μου. Πολύ σύντομα να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Ευχαριστούμε κύριε Άντερ. Ο κύριος Καρβαλό, εκ μέρους της Επιτροπής. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο και να αναφερθώ σε μία σημείο στα σχόλια που έγιναν. Πρώτον, ευχαριστούμε την κυρία Μέρκης η έκθεσή της αποτελεί μια πολύ καλή βάση για γνωμοδότηση. Αρχικά θέλω να πω ότι η ανακοίνωσή μας για τις πρώτες ύλες καλύπτει όχι μόνο τα ορυκτά, αλλά και αυτό που εσείς ε, αναφέρατε ως βιωτικούς πόρους. Για παράδειγμα, καλύπτει και το ξύλο και τα ελαστικά. Ε, στην Επιτροπή έχουμε τρεις πυλώνες. Εδώ πέρα αυτό που αναφέρεται είναι αυτό που εμείς θεωρούμε ως τρίτον πυλώνα, ε, αποδοτική χρήση και ανακύκλωση των πρώτων υλών. Δεν υπάρχει μια προτεραιότητα στους, στους, πυλώνες, όλοι είναι ίσως, ε, εξίσου σημαντικοί. Φτάνω στο σημείο 2 το ζήτημα των στόχων. Εμείς συμφωνούμε με τις απόψεις ε, ε, που εκφράστηκαν εδώ για την δυσκολία θέσης ενός, προσδιορισμού ενός αριθμητικού στόχου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε υπέρ της αποδοτικότητας ε, των πρώτων υλών. Η Επιτροπή βεβαίως συμφωνεί και έχει υιοθετήσει, έχει κάνει μια ανακοίνωση για εμβληματική πρωτοβουλία. Αυτή τη στιγμή συντάσσουμε και ένα οδικό χάρτη. Το θέμα είναι, έχουμε την απαραίτητη μεθοδολογία για να το εξετάσουμε. Μήπως είναι καλύτερο να τα εξετάσουμε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση της ανακύκλωσης, για παράδειγμα, πρόσφατα η Επιτροπή στην Οδηγία για τα Απόβλητα έθεσε ορισμένους στόχους ε, για την ε, ανακύκλωση αλλά σε συγκεκριμένε περιπτώσεις. Μήπως μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε κατά περίπτωση όταν αυτό είναι ρεαλιστικό. Για να μην δημιουργήσουμε έναν πυρετό, αν θέλετε, που δεν θα είναι ρεαλιστικό. Στο σημείο 6 αναφέρεστε στο, ζήτημα, στο ένα σύστημα καταγραφής της, ε, ε, της προέλευσης των πρώτων υλών αλλά δεν κατανοούμε ακριβώς ε, τι εννοείται. Στο, το flagged, για παράδειγμα, που αναφέρεται, ε, σχετίζεται με τα δάση. Μπορούμε να δούμε ορισμένε ορισμένες δυνατότητες, αλλά όχι πάντα, σε ορισμένες περιπτώσεις. Στο σημείο 9 αναφέρεστε ε, στα ορυκτά που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες. Δεν έχουμε θέση, ε, λάβει μια οριστική θέση. Κατά τη γνώμη μας, είναι καλύτερο να τα εξετάζουμε ε, αυτά τα ζητήματα κατά περίπτωση και όχι γενικά. Σημείο 8. Το ζήτημα της βιοπικιλότητας ε, και της συμφιλίωσης ε, οικονομίας και περιβάλλοντος. Αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Και πάλι να πω ότι πέρσι δημοσιεύσαμε ορισμένες κατευθυντήρες γραμμές για το Natura 2000 στοχεύοντας ειδικά σε αυτή την ε, παροχή καθοδήγησης, αν θέλετε, προς τα κράτη-μέλη και στις τοπικές αρχές για το πώς να συμφιλώσουν αυτά τα δύο διαφορετικά περιβάλλοντα. Δεν ξέρω αν μένουν πολλά ακόμα να γίνουν. Τέλος, σημείο 11. Αναφερθήκατε στους ορυκτούς πόρους και τους, και τους φόρους επί αυτών των ε, ε, πόρων. η δημιουργία ενός φόρου που δημιουργεί με τη σειρά του κόστος που το οποίο δεν επομίζονται οι εξωτερικοί ανταγωνιστές, αυτό ε, δημιουργεί μειονέκτημα για την ε, οικονομία μας. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, υπάρχει δυνατότητα ε, μεταφοράς ενός φόρου από την εργασία, από την απασχόληση στους, στις πρώτες ύλες. Αν ο γενικός αντίκτυπος δεν είναι υψηλός, σε επίπεδο κόστους, να το εξετάσουμε. Αυτό το ζήτημα απαιτεί οικονομική ανάλυση. Αλλά θα ήταν χρήσιμο να το κοιτάξουμε. Το τελευταίο μου σχόλιο. Κάποιος είπε τι εργαλεία και μέσα μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να είμαστε πιο αποδοτικοί. Ε, στην αξιοποίηση των πρώτων υλών, των φυσικών πόρων και ε, στην ανακύκλωση. Εδώ υπάρχει μια θετική απάντηση από την κυρία Μέρκης για άμεση εφαρμογή των εταιρικών σχέσεων καινοτομία. Όπως ξέρετε, αυτό ε, συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή προετοιμάζει μια πρόταση για την, ε, τις εταιρικές σχέσεις για τους φυσικούς αυτούς πόρους. Και εμεί θεωρούμε ότι αν θέλουμε να σημειωθεί πρόοδο, πρέπει να υπάρχει μια δομή των συζητήσεων με τα κράτη-μέλη, το κοινοβούλιο, τους, ε, τα ενδιαφέροντα μέρη. Και όλα αυτά τα ζητήματα που μα αφορούν σήμερα θα τα εξετάζουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Έχουμε την απαιτούμενη τεχνολογία για να επιτύχουμε αυτή την ενεργειακή αποδοτικότητα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, πρότυπα, ε, ε, για τις δημόσιες προμήθειες. Υπάρχουν πολλές τέτοιες πτυχές. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητούμε ε, συχνά, ανατακτά διαστήματα και ιδιαίτερα να δούμε αν όλα αυτά είναι εφικτά. Το να έχουμε μια συζήτηση μια φορά το χρόνο, μια φορά τα δύο χρόνια, δεν αλλάζει κάτι. Γιατί κατά τη γνώμη μου επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Μια εταιρική σχέση καινοτομία λοιπόν μπορεί να αποτελέσει μια λύση για την ύπραξη συστηματικού διαλόγου για όλα αυτά τα ζητήματα. Ε, μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένου στόχου, σε ποιο πράγμα και μέχρι πότε. Με ποια προθεσμία. Δηλαδή από τι γενικόλογε γενικόλογες μπορούμε να περάσουμε στα αυτά αποτελέσματα. Κρίσιμη σημασία σε αυτά τα ζητήματα αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε μια δομή, να διαρθρώσουμε αυτόν τον διάλογο, κάτι που δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις σας. Αν ήθελε ε, η συγγήτρια να προσθέσει κάτι. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ. Αρχικά σας ευχαριστώ για τις ε, επικοδομητικές σας παρατηρήσεις, αλλά και για τις φιλοφρονήσεις σας. Πολύ σύντομα. Έχουν ε, αναφερθεί πολλά ερωτήματα. Θα απαντήσω κυρίως στα ερωτήματα. Θα πρέπει βεβαίως να το εξετάσουμε ενδεχομένω ε, μαζί ε, ορισμένα σημεία, δηλαδή που χρειάζονται, χρήζουν περαιτέρω εξήγηση. Γι' αυτό που ανέφερε ο κύριος Φλόρενς. Πράγματι, δεν μπορούμε να θέσουμε μόνο στόχους, αλλά πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι, αναφέρθηκε ως ε, case by case κατά περίπτωση εξέταση. Δηλαδή, ο προσδιορισμός στόχων δεν, δεν, είναι, δεν είναι σκόπιμος. Με την ανακύκλωση πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς. Όχι δηλαδή 17% ή 70% έχει ανακυκλωθεί, αλλά τι ακριβώς παράγουμε από αυτή τη διαδικασία. Εκεί, για παράδειγμα, η ανακύκλωση θα πρέπει να ε, χωρίζεται σε τρία στάδια. Ε, η συλλογή, του υλικού, η προεπεξεργασία ή διαχωρισμός και μετά refinery smelting. Έχουμε λοιπόν τρεις ε, ξεχωριστές φάσεις και τα το, περισσό, το μεγαλύτερο μέρος του υλικού διαχωρίζεται εκεί. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο ακριβείς λοιπόν εδώ. Στη συνέχεια, η ιεράρχηση που ανέφερα για τις πρώτες ύλες. Δεν λέω ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτό. Λέω απλώ ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι οι πρώτε ύλε μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικού τρόπου ε, και δεν χρησιμοποιούνται πάντα με τον ε, πλέον κατάλληλο τρόπο. Επειδή ακριβώς έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ διαφόρων υλών και τρόπων αξιοποίησης, θα πρέπει να το εξετάσουμε περισσότερο αυτό. Ε, αναφέρθηκαν οι ανεμογεννήτριες Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν ορισμένα υποκατάστατα για το δικό σας παράδειγμα. Και πάλι, δεν λέω ότι πρέπει να σταματήσει αυτό, απλώς θα πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Για τον φόρο τώρα, πολλά υπόθηκαν εδώ. Στόχο μου δεν είναι να συσσωρεύσουμε φόρους, αλλά Βεβαίω, ε, λέμε ποια είναι τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Ακριβώ, τα δημοσιονομικά ε, εργαλεία είναι πολύ σημαντικά για να ενθαρρύνουμε ε, μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Και είναι σημαντικό να εξετάσουμε αυτή την μεταφορά φόρου από την απασχόληση στην ε, φορολόγηση πρώτων υλών. Για παράδειγμα, αν η απασχόληση γίνει πιο φτηνή, πολλά μπορούν να διορθωθούν, ε, να επισκευαστούν. Γιατί πολλοί προτιμούν να αγοράσουν κάτι καινούριο από ότι να το επισκευάσουν. Τώρα για τον συνάδελφο κύριο Γερμπράντη. Πολύ σημαντική η βιοπικιλότητα, συμφωνώ μαζί σας και θα πρέπει να, το να έχουμε μια ολοκληρωμένη ε, πολιτική γι' αυτό. Όχι δηλαδή κατακαιρματισμένα πρώτα να κοιτάζουμε την βιοπικιλότητα μετά τις, ε, ε, τους φυσικούς πόρους και το καθεξής. Μία και μόνο στρατηγική θα πρέπει να υπάρχει για αυτά τα σημεία. Όχι μια κατακρεματισμένη πολιτική επειδή έχουμε 20 διαφορετικούς επιτρόπους. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αυτό κάποια στιγμή. Μετά. Για την εφαρμογή. Πράγματι, πολύ συχνά, όταν θέλουμε κάτι πολύ, δημιουργούμε νέα νομοθεσία. Και έτσι προσθέτουμε περισσότερα, ακόμα περισσότερες νομικές πράξεις. Γι' αυτό και εμείς εστιάζουμε ιδιαίτερα στην εφαρμογή. Ας φροντίσουμε δηλαδή το οικοδόμημα που έχουμε από ότι να φτιάξουμε μια νέα πτέρυγα. Διακόπτη, Πρόεδρος, δυστυχώς θα πρέπει να σας ζητήσω να ε, ολοκληρώσετε. Έχω ακόμα ε, ορισμένες ερωτήσεις που έχουν τεθεί. Κύριε Άντερ, Πρόεδρος, δεν θα υπάρξει διερμηνία. Θα σταματήσει η διερμηνία. Τότε να ολοκληρώσω τα αγγλικά. Εφόσον δεν θα έχουμε διερμηνία. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές, αλλά ε, ιδιαίτερα για τους φόρους ε, και τα λοιπά. Και τέλος, ε, για την εταιρική σχέση καινοτομίας που ανέφερε η Επιτροπή, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε δει ακόμα το περιεχόμενο αυτής της εταιρικής σχέσης καινοτομίας. Θα ήθελα να, την, να το δω αυτό το περιεχόμενο, θα ήθελα να στηρίξω αυτή την ιδέα, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι περιλαμβάνει η πρότασή σας. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας εξηγήσετε περισσότερο, περαιτέρω στις επόμενες ε, συνεδριάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τις διερμηνείς. Οι τροπολογίες πρέπει να υποβληθούν ε, μέχρι τις 27 Μαΐου ε, στις 12 η ώρα.